je vous propose de euh, reprendre vos échanges de souvenirs de vacances après la réunion. Καλή σας μέρα. Ας ε, προτείνω να ξεκινήσουμε. Ε, πρώτη συνεργασία μας μετά τις διακοπές. Ελπίζω να περάσατε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλή επάνωδο. Με μια ημερήσια διάταξη φορτωμένη. Σε ό,τι αφορά την έγκριση μερίσιας διάταξης, να σας πω ότι θα τροποποιηθεί ως εξής. Το σημείο 12, ε, έκθεση Παπαδοπούλου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα σπουδές ανταλλαγέ μαθητών, την έμιστη άμιστη κατάρτιση, την εθελοντική εργασία και την απασχόληση ω εσωτερική άμιστη βοηθή. Αυτό θα πάει πριν το σημείο 10 έκθεση Bauer για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Το 12 λοιπόν μετακινείται πριν το 10, αν δεν, αν δεν έχετε αντίρρηση. Οι συγκεκριτές δεν είναι εδώ, αλλά ε, γνωρίζω ότι συμφωνούν. Αποφασίστηκε. Σημείο 2. ανακοινώσει τη Προέδρου. Έξι ανακοινώσει. Πρώτον. Σε ό,τι αφορά την τελική έκθεση της Επιτροπής ε, Προπολογισμών για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θυμάστε ότι η Επιτροπή μας είχε εκφέρει γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αρχή της διαδικασίας. Οπότε το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να υποβάλουμε μια καινούρια ε, γνωμοδότηση. Όμως η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα υιοθετήσει τη δική της σύσταση στο τέλος των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε η Επιτροπή Απασχόλησης, όπως και οι υπόλοιπε επιτροπές οι οποίες είχαν ήδη εκφέρει γνώμη παλαιότερα, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ε, υιοθετήσουν καινούργια γνωμοδότηση. Πολύ περισσότερο που η Επιτροπή Προπολογισμών θα πει στη γνωμοδότηση αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μόνο. Σας θυμίζω ότι το θέμα το οποίο είχε προβλεφθεί να εγγραφεί στην μέση διαταξή της ε, Τρίτης ε, θα αναβληθεί. Το ίδιο και η ψηφοφορία. Θα αναβληθούν για την σύνοδο, τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου όταν πλέον θα είναι έτοιμο το μεγαλύτερο τμήμα της νομικής βάσης. Για μας αυτό αφορά προφανώς την ε, έκθεση Γιούτα Steinbrück ε, το κωδικό όνομα είναι easy πλέον και όχι ψή και ελπίζουμε να έχουμε έτοιμα και δύο άλλα ζητήματα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι μπλοκαρισμένο στην, ε, στο Συμβούλιο το των Απόρων. Ε, γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι θα είναι έτοιμο στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. χρειάζεται να δούμε ποιες είναι οι ελάχιστες συνθήκες που θα μας βοηθήσουν να το ξεμπλοκάρουμε. Η έκθεση αυτή εδώ στην Επιτροπή είχε εξασφαλίσει μεγάλη πλειοψηφία, το ίδιο και στην Ολομέλεια. Αυτό το υπενθύμησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στην ομάδα επαφής χτες. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό το ζήτημα αυτό για το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεμπλοκάρουμε. Δεύτερο σημείο. Διάσκεψη που οργανώνουμε εμείς με τις τέσσερις υπηρεσίες που βρίσκονται στην ευθύνη μας. Όπως το κάναμε και τον Ιούνιο του 2011. Οργανώνουμε αυτή τη διάσκεψη ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο, αποφασιστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας. θα εστιάσουμε στο πώς μπορούν οι τέσσερις υπηρεσίες να βοηθήσουν. Θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου από τις 9.30 ως τη 1 και η δική μας διάσκεψη θα γίνει το απόγευμα και την επόμενη μέρα. Και η δική μας συνεδρία θα γίνει το απόγευμα και την επόμενη μέρα. Το πρόγραμμα θα διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα. Σας καλώ να συμμετάσχετε ε, μαζικά. Επίσης, να σας πω ότι δεν ακυρώθηκε καμία διερμηνία, οπότε έχουμε βελτιστοποιήσει τη χρήση του υπερπολογισμού μας. Τέταρτη ανακοίνωσή μας, η εξέλιξη του θέματος του, του χρόνου FLG, Flight, Flight Time Limitation, περιορισμού του χρόνου πτήση. Η... ιδιαίτερος ε, το, τους πραγματικ, τις πραγματικές συνθήκες εργασίας όχι μόνο των πιλότων αλλά και όλου του προσωπικού αέρος στον τομέα των εναέριων μεταφορών συνδικαλιστές ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως. Η Επιτροπή Μεταφορών βέβαια είναι ε, υπεύθυνη της ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε την επιτροπολογία για αυτό το ζήτημα σύμφωνα με τις συστάσεις της ε, ΕΖΑ. Εμείς από τη δική μας πλευρά ε, οργανώσαμε μία ε, ακρόαση ε, ρώτησα τους ε, εισηγητές και συμφώνησαν ε, να έλθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Μεταφορών εντός των προθεσμιών και να τους πούμε ότι έχουμε αμφιβολίες για την ικανότητα του Κοινοβουλίου να εγκρίνει αυτή την, την, τη διαδικασία επιτροπολογίας και θα προσφύγουμε και στην νομική υπηρεσία για να διαπιστώσουμε αν Πράγματι, πρόκειται μόνο για θέματα μεταφορών. Ε, οι συνδικαλιστές απευθύνονται σε εσά με email λέγοντας ότι ε, δεν ζητήθηκε η γνώμη τους από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Ε, μην, ας έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Τα συνδικάτα ενδεχομένως τυπικά είπαν τη γνώμη τους Έγινε κάποιος ε, διάλογος. Αυτό όμως που δεν πέρασε είναι το μήνυμά τους. αυτή την έννοια λοιπόν δεν ακούστηκαν. Δεν ακούστηκε η φωνή τους και γι' αυτό το λόγο απευθύνονται σε μας. Ε, η Ευρωπαϊκή του Ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο δεδομένης της, ε, του ευαίσθητου του θέματος, δεδομένου του ευαίσθητου θέματος θα πρέπει να το δούμε και μας απασχολεί όλους. Επόμενο ζήτημα. Η Κριστίνα και η Λάρα ε, πέρασαν στη γραμματεία της Επιτροπής μας από Σεπτεμβρίου ως βοηθή. Δεν είναι εδώ. Θα τις παρουσιάσουμε όταν έρθουν, όταν τις βρούμε. Θα έπρεπε να έχουμε βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Τέλος πάντων, σίγουρα είναι πολύ Ε, Έκτη ανακοίνωση, ε, η συνεδρίαση μας μεταδίδεται μέσω ίντερνετ. Ε, σημείο 3, ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Alors, le rapporteur du point 3 n'étant pas là, je vous propose... Οπότε, σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 4. ο λόγος στη Μαρίαν Χάρκιν. Διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε έναν ε, άτυπο τριμερή διάλογο και καταλήξαμε σε προσωρινή συμφωνία καταρχάς για το ειδικό καθεστώς για τη γεωργία και δεύτερον για τους στόχους και το πεδίο ώστε να καλύψουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και από την παγκοσμιοποίηση και από την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλέ φορέ απευθύνει έκκληση προ το σκοπό αυτό. Κάποια τεχνικά ζητήματα έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί προσωρινά Αυτά αφορούν κριτήρια παρέμβασης άρθρο 4, συμπληρωματικότητα, συντονισμό άρθρο 9, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών άρθρο 10, ε, ενημέρωση πληροφόρηση δημοσιότητα 12, ε, ρεσιμότητα 15, προϋπολογισμός 10, 15, διαχείριση του προϋπολογισμού 21, απόδοση εισφορών 22, και όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται πως έχουν κλείσει, αλλά δεν έχουν κλείσει ακόμα πολλά και σημαντικά θέματα. Από τα εκκρεμή λοιπόν σημαντικά θέματα έχουμε μία πρόταση του Συμβουλίου για συμπερίληψη των νέων από 15 έως 24 ετών, μια τελείως νέα πρόταση, η οποία ε, ενεργοποιείται όταν ένα κράτος μέλος καταβάλει αίτηση, καταθέσει αίτηση για ε, υποστήριξη ανέργων από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης ακόμα και αν στηρίζονται, στηρίζεται το κράτος μέλος αυτό και από το Ταμείο για την Αντιμετώπιση Ενέργειας, ε, το νέων πάλι μπορεί να ζητήσει α, τη χρηματοδότηση αντίστοιχο αριθμό για τις ηλικίε 15-24 ετών. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός του πεδίου του κανονισμού, αλλά πάντως εξετάζουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Καινούρια πρόταση, όπως είπα. Επίσης, έχουμε κάποια εκκρεμή ζητήματα ως προς τον προσδορισμό του ποιος είναι ο εργαζόμενος. Εάν απαιτείται να περιοριστεί στους μονίμως εργαζομένους, ε, στις άλλες μορφές απασχόλησης, Έχουμε επίσης τα ζητήματα των, των ε, ποσοστών συγχρηματοδότησης που όπως ξέρετε έχει αποφασιστεί μια διαβάθμιση της συγχρηματοδότησης ανάλογα με το κράτος μέλος, την κατάστασή του, την οικονομική δηλαδή, αλλά από την πλευρά του Συμβουλίου έχει προταθεί μια πάγια αναλογία αναλογής 50 50-50 Επίσης ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία και πιστεύω θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε θα είναι οι προσωποποιημένες υπηρεσίες και το ποσοστό της χρηματοδότησης που μπορεί σε αυτές να χορηγηθεί. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιδότηση κινητικότητας, γενικά ενισχύσεις υπό τον τίτλο των προσωποποιημένων υπηρεσιών. Ο προσεχής άτυπος τριμερής διάλογος είναι σήμερα και προβλέπεται ακόμη μια σειρά τριών τριμερών διαλόγων. Πιστεύω ότι παραμένουν αυτά τα θέματα εκρεμή και όπως γνωρίζετε έχουμε περάσει ήδη πολύ καιρό περιμένοντας απόφαση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και για δίποτε ασχετική πρόταση από πλευρά του Συμβουλίου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα ήμασταν τυχεροί εάν μέσα στους τρεις προσεχείς ε, τριμερείς διαλόγους μπορέσουμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητες. Μήπως κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο, Φρεντήρικ Ντάρντεν. Δύο λογάκια. Επιβεβαιώνω τα όσα μας είπε η συγγήτρια για τις διαπραγματεύσεις ε, και η Προεδρία του Συμβουλίου ακριβώς έχει μια παράξενη, πολύ παράξενη στάση έτσι, και το Συμβούλιο δεν θέλει να κινηθεί ουσιαστικά και δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο θα αναλάβει τις ευθύνες του γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα δύσκολα προς ρύθμιση. και σύμφωνα με τον ορισμό του εργαζόμενου ακριβώς ε, εντάξει θα το δούμε αυτό και η συγχρηματοδότηση πρόκειται για πιστοδρόμηση από πλευρά Συμβουλίου και χρειάζεται να το προσέχουμε και για τους νέους τώρα μια πρόταση που ίσως είναι ιδιαίτερα ελκυστική έχουμε μια χρηματοδότηση από το Αρμόδιο Ταμείο και για τους νέους άνεργους αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει δεν στέκει εκεί και είναι και κάτι το υποκειμενικό. Γι' αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Το Συμβούλιο όμως πίεση ασκεί σχετικά με αυτό το σημείο. Θα πρέπει να δείξουμε πρωτοτυπία για μια λύση και για τα μέτρα που θα επιλέξει κανείς. Προσέχουμε σμένα πράγματα και δεν τα διατηρεί το Συμβούλιο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι να αναλάβουν τον τομέα αυτό και θα πρέπει να το επιμείνουμε ώστε να διατηρηθεί. Ευχαριστώ. Ναι, λέει πρόεδρος. Μήπως κάποιος άλλος θα επιθυμούσε το λόγο τώρα. Όχι, κανείς. Ε, υπεύθυν ε, για την ομάδα διαπραγματεύσεων ε, ευχαριστήσω πήραν το λόγο και όσα είπαν και για το Κοινοβούλιο στη φάση αυτή για να δεχτούμε τις όρους της πολιτικής συμφωνίας στο Συμβούλιο και πρόκειται για την επιβίωση του Ταμείου αυτού της προσαρμογής ε, για την παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι το αντίτιμο, αυτές οι διατάξεις, οι ρυθμίσεις ε, εντάξει είναι κάπως ε, τρελές τρελές αλλά είναι μια νομική βάση όμως και να μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν για την απασχόληση νέων και είναι και ένας κίνδυνος παράκαμψης του θέματος και χρειάζεται κανείς να πληρεί τις προϋποθέσεις όμως τις νέες οι οποίες τίθενται, ορίζονται και το να μπερδευτούν οι νομικές βάσεις ε, αυτό δημιουργεί σύγχυση και όλη η διαχείριση περιπλέκεται και στη συνέχεια δεν μπορεί κανείς ε, να καταλάβει ποιο είναι το αντικείμενο, τι αφορά κάθε ταμείο, που η Επιτροπή εδώ έχει την ε, αρμοδιότητα. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, το έκανα ήδη στην ομάδα διαπραγματεύσεων. Θα το επαναλάβω όμως εδώ. Και στο Συμβούλιο υπάρχει μια διάθεση βέβαια για πολιτικές ενδείξεις υπέρ της απασχόλησης νέων και εμείς δεν θέλουμε να μειονεκτήσουμε απέναντι σε αυτό το θέμα, χρειάζεται να είναι προτεραιότητα, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις και θα πρέπει να δούμε το αντικείμενο αυτού του ταμείου και με την εισηγήτρια είναι από τα σημεία πάνω στο οποίο είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε πραγματικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι τελειώσαμε έτσι με το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Μενράιτεν που θα αντικαταστήσει τον κύριο Τσαμπάουρη που αδυνατεί να αδυνατούσε να προσέλθει. Άρα λοιπόν να μας πει μερικά πράγματα για το σημείο 3 για το γενικό Μισό λεπτό, μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος να κοιτάξω κάτι για να μας παρουσιάσει μάλλον ε, τις τροπολογίες για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 και που αφορά όλα τα τμήματα. Οι τροπολογίες είναι 65 από τους συναδέλφους πάνω σε σου και 12 για τα υπόλοιπα. Κυρία Ομενρό ήταν, έχει το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για να σας πω κάτι ότι σήμερα το πρωί δεν μπορούσε κανείς να περάσει, υπήρχε τρομερή κίνηση στους δρόμους, γι' αυτό και η καθυστέρηση. Κυρία Πρόεδρε, όνομα του συναδέλφου θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ, προσέξτε με. Ο εισηγητής έχει διαφορετική άποψη από τον εισηγητή της σοσιαλιστικής ομάδας. Το πρώτο σημείο αφορά το προσωπικό προσωρινό, με προσωρινό συμβόλαιο, αλλά και τους μόνιμους υπαλλήλου ε, με μία μείωση 5% του προσωπικού. Είμαστε κατά της τροπολογίας αυτής. Το ίδιο ισχύει και για το 6547 και για το 6560. Είμαστε κατά και του 65-62 διότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο μικρό πρόβλημα, στο αποκαλέσουμε έτσι. Και το 65-09 που αναφέρεται ο κοινωνικός διάλογος που θέλει στο ιδιοκιούπι να βάλει επιτροπή. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες του συγητή πάνω στο θέμα αυτό και ελπίζουμε το ίδιο να πράξουν και οι υπόλοιποι. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Μισό λεπτό, να κοιτάξω τα χαρτιά μου. Το 040303 πρωτοβουλία για τους νέους. Θα ήθελα να πω το εξή ότι για τη φιλελεύθερη ομάδα δεν είναι για την αύξηση του ποσού. Δεν πρόκειται για κάτι τι, αλλά για να έχουμε ένα extra front loading ώστε οι πρωτοβουλίες αυτές που αναλαμβάνονται στο σχετικό τομέα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω 1,7 εκατομμύρια αντί για 1,5 εκατομμύρια ένα extra front loading, ένα πλέον ποσό που θα αφιερωθεί σε αυτό λοιπόν. Και ακόμη κάτι. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Το σχέδιο πιλότο για το benefit scheme. Η ομάδα μου στην προπαρασκευαστική συνάντηση υποστήριξε αντιμετωπίζει προβλήματα για το θέμα αυτό. Γιατί οι διάφορες οργανώσεις δεν χαίρονται και πολύ για τα όσα εμείς θα επιθυμούσαμε να κάνουμε και πώς ε, ξεκινώντας από την Ευρώπη θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πραγματικά την ε, εξέβρεση θέσεων εργασίας, να βοηθήσουμε τους άνεργους. Και τα ποσά που απαιτείται να εξευρεθούν θα πρέπει να πληρωθούν στα κράτη-μέλη σχετικά και με την φορολόγησή τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν τα συζητήσαμε και τόσο χθες, αλλά δεν νομίζουμε ότι σχετικά με το θέμα αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, επιδοτήσεις. Η θέση του εισηγητού πάντως ε, είναι γνωστή σε όλους, ε, έχει αποσταλεί. Ευχαριστώ πολύ. Νταχντάν. Πολύ σύντομα δύο λόγια, Πρόεδρε και θα μιλήσω τρία θέματα, τρία σημεία. Καταρχάς την έκθεση του κυρίου Ορή που έχουμε καταθέσει τροπολογίες επιμένοντας κυρίως ως προς την αναγκαιότητα για ένα κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο για την κοινωνική πολιτική και προκειμένου διατυπώνουμε τη λύπη μας για τον περιορισμό στον τίτλο 1β. Επίσης θέλουμε να ενισχυθούν τα ποσά για την εγγύηση νεότητας και να δοθούν επιπλέον εγγύησεις για τα προγράμματα πρόοδος, ωρές και ταμείο προσαρμογής. Ε, επίσης, έχουμε καταθέσει τροπολογίες για να ενισχύσουμε το σχέδιο του προπολογισμού της Επιτροπής και υποστηρίζουμε και άλλες τροπολογίες ε, που ζητούν περισσότερο από ό,τι οι μας ε, την ενίσχυση του Κοινωνικού Ταμείου, Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, υποστήριξη των ε, για την αντιμετώπιση τη φτώχεια κτλ στις προπαρασκευαστικές δράσεις. Υποστηρίζουμε βεβαίως τα έργα τα οποία έχουν κριθεί ως πιο σημαντικά, έχει δοθεί βαθμός προτεραιότητας υψηλός δηλαδή, και βέβαια το θέμα της, ε, του επιδόματος ανεργίας, του ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας ε, και την ενίσχυση των νέων και ιδιαίτερα την κινητικότητα. Ευχαριστώ πολύ, δεν περίμενα ότι θα συζητούσαμε το θέμα αυτό τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι πριν την ψηφοφορία θα, θα έπρεπε να γίνει συζήτηση του άλλους. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή συνεπή μετά όσα έχουμε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ακολουθήσει όλο το προηγούμενο έτος και γι' αυτό προτείνουμε με να γίνει αποδεκτή αυτή η γραμμή του προπολογισμού, αλλά θέλουμε υψηλό επίπεδο δαπανών στους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη ευθέω, πράγμα το οποίο όμως θα σημαίνει ταυτόχρονα περιορισμό των δαπανών σε κάποιους άλλους τομείς. Δεν θέλουμε λοιπόν να εμφανιζόμαστε φάσκοντες και αντιφάσκοντες. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε τη λύπη μας γιατί την κάποιων δαπανών, τις οποίες έχουμε ζητήσει για να ενισχύσουμε κάποιου άλλου τομείς υποδομές κτλ. Και έτσι ο δικός μας ο κατάλογος ψηφοφοριών με κύριο μέλημα πάντα τη συνέπεια Υποστηρίζει βέβαια την ε, εγγύηση για τους νέους μικρές ε, αυξήσεις στην ε, χρηματοδότηση κάποιων τομέων και θα τις υποστηρίξουμε αυτές. Αλλά δεν έχουμε βάλει θετικό πρόσημο σε ένα ε, σύστημα ευρωπαϊκό επιδόματος ανέργειας. Και ως εκ τούτου, αφού δεν υποστηρίζουμε την ιδέα την ίδια, δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε και τη σχετική χρηματοδότηση. Πάντως, εν γέννη, είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των τομέων εκείνων του προπολογισμού που μπορούν να δώσουν όθηση ουσιαστική στην ανάπτυξη. Και άρα άλλους τομείς, όσο και να θέλαμε, δεν μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Για την τροπολογία 65-16, ε, την οποία ανέφερε κύριε Ρόιτεν, η ιδέα υποστήριξε αυτή, αυτού του σχεδίου πιλότου με μια ε, μελέτη της Κομισιόν, δηλαδή να υποστηρίξουμε αυτή τη μελέτη που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν, υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, ελάχιστου επιδόματος ανεργίας. Ε, αυτό το σημείο συμφωνήθηκε από τους συντονιστές του ΕΛ και των Σοσιαλιστών ως σημείο προτεραιότητας μεταξύ των πιλωτικών σχεδίων που θα ε, υποστηρίξουμε. Η, γνώμη του συγητή είναι θετική Και ε, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της ακρόασης, πολύ σημαντικής ακρόασης που οργανώσαμε τον Ιούλιο, θα ε, επέτρεπε αυτή η απόφαση να γίνει η μελέτη, να διενεργηθεί μια τέτοια μελέτη, που, κάτι που θα ξεπερνούσε κατά πολύ τις ε, ε διαπραγματεύσεις με τους συνδικαλιστές, λαμβάνοντας υπόψη όμως τη γνώμη τους, τίθεται ένα θέμα ισορροπίας μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης και ε, ενδεχομένως θα επέτρεπε ένα τέτοιο σύστημα να μειώσει αυτές τις ανισορροπίες. Ε, η Κομισιόν ε, θέλει να κάνει μια τέτοια μελέτη, να ξεκινήσει να δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε τμήμα της διαπραγμάτευσης, έχουμε συμφέρον να ε, βάλουμε και εμείς το χεράκι μας έτσι ώστε να μην αφήσουμε μόνο ε, τους υπεύθυνους των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ θερμή ε, υπέρ της υποστήριξης ε, του, σχεδίου πιλότ, του πιλωτικού σχεδίου. Σας υπενθυμίζω ότι σοσιαλιστές και ΕΛΚ συμφώνησαν, τώρα από εκεί πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Τελειώσαμε αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξης και περνάμε στις πιοφορίες. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τις ε, ε, κάρτες μας. Μπορούμε, μπορούμε όμως να δούμε... Α, αν βάλετε τις κάρτες σας να δούμε αν δουλεύουν τα μηχανήματα και να δούμε ποιος την έχει και ποιος την έχει ξεχάσει. Όλοι έχετε τις κάρτες σας, ο αριθμός είναι σωστός. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5. Ξεκινάμε με... Alors, 5, ε, Σημείο 5. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014. Όλα τα τμήματα. Ψηφίζουμε καταρχήν τα νούμερα. Μηδέν τέσσερα, μηδέν Τροπολογία 67, 47 υπέρ κατά αποχές. Συγγνώμη, 65-47. Ε, τροπολογία του εισηγητή 6.500. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, εξωτερικό προσωπικό, τροπολογία 65-48. Φρεντερικ Ταρντέν, υπέρ. Φωτογράφοι με εμποδίζουν λίγο. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 65-60 της κυρίας Ζούμπερ. Ε, για το κοινωνικό ταμείο υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Για το ίδιο θέμα 65-01 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, μετά για το ψι που έγινε easy αργότερα. Ε, τροπολογία 6502 και 6544 είναι οι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνεται. Για το κοινωνικό ταμείο και πάλι περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, δύο ταυτόσιμες τροπολογίες εισηγητή και νταρντέν, 6503-6550 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, περιοχές 6504 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάλι κοινωνικό ταμείο ε, τροπολογία 6505 του εισηγητή και 6551 του κ. Νταρντέν. Όχι, καταρχήν του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6551 καταπίπτει. Και πάλι για τις μειοκτούς περιοχές, 6506 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6552 πίπτη. Τώρα περνάμε για την πρωτοβουλία για την αποσχόληση των νέων. Τροπολογία 6561 της κυρίας Σούμπερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία τα του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τροπολογία 65-62 της κυρίας Σούβερ. η συγγήτρια είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 1 για τον κοινωνικό διάλογο. Συγχετρία είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, α, εγκρίνεται. Περνάμε στη σελίδα 6, ε. ε. Nous en euh, Σελίδα 7, τροπολογία 65-36 του εισηγητή. Ανάλυση και ε, μελέτης για την κοινωνική κατάσταση, τη δημογραφία και την οικογένεια. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65-08 του εισηγητή. Για το progress υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 6508. Κλείνει η ψηφοφορία. 17 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65-35 του εισηγητή. Νομίζω ότι αφορά το ίδιο ζήτημα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65, 46 και 65, 63 καταπίπτουν. Περνάμε στην 65, 25 του εισηγητή για το πράγμα Γιούρες με προφορική τροπολογία κατόπιν αιτήματος της ομάδας φιλελευθέρων. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65-26 καταπίπτει, το ίδιο και 65-49. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και μικροχρηματοδοτήσεις, 65-28 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 65, 34, 65, 53 και 65, 64 καταπίπτουν. Περνάμε στην τροπολογία 65-38 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στο Ίδρυμα για την Βελτίωση των ε, Συνθήκων Εργασίας και Ζωής. 6527 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρινεται 6554 65-54 κατά πίπτη. Τώρα 5 για, την, ε, για το Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας στην Ασία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο για την ολοκλήρωση του Progress 6531 και 6557 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο και για το Eures 6532 και 6556 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για τις άλλες δραστηριότητε και πάλι το ίδιο, 65, 33 και 65, είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, δράση προετοιμασίας, ε, το κέντρο πληροφορίας, ε, πληροφοριών 65-41 της κυρίας Στάινρουκ και της Γιούτα Χάουκ καταπίπτει λέει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 Ce 65-13, il vient après. C'est pas. Alors, euh, il y a une erreur sur le commentaire. Υπάρχει ένα λάθος στο κείμενο, στα σχόλια. Δεν έχουμε ψηφίσει την 65-13. Οπότε η 65-40 έπρεπε να ψηφιστεί ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. 65-13. Νομίζω ότι απορρίπτεται, ας το επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 6541. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. 30 υπέρ, 5 κατά, 2 εποχές. Εγκρίνεται. Δύο επόμενε τροπολογίε καταπίπτουν. Φτάνουμε στην 65 του εισηγητή ε, για την απασχόληση των νέων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65-66 καταπίπτει. Πιλωτικό σχέδιο για την προσθέμενη εξένωση ε, συστήματος συστήματο ευρωπαϊκών επιδομάτων ανεργία. Τροπολογία 65-16 υπέρ. Κατά. Πρόκειται για την 6516. Οι συντονιστές του ΕΛΚ ήταν υπέρ όταν το συζητήσαμε στην άντληση των συντονιστών. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 6516. Tout le monde a pu voter Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή. Εγκρίθηκε. 65-17. Ήταν το πιλωτικό σχέδιο για την ε, αποφυγή των διακρίσεων. Η τροπολογία του εισηγητή εκ μέρους τη Επιτροπή Απασχόληση. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 65-18 τροπολογία του εισηγητή για το πιλωτικό σχέδιο για το, την κοινωνική Υπέρκατα κατά αποχές 6540. 65-40 προπαρασκευαστική ενέργεια. Για να δούμε, για να δούμε. Ε, κοινωνική επιχειρηματικότητα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65-19 τροπολογία για το Ταμείο Αυτοπροσαρμογής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65-20-65-59 ταυτόσημες ψηφίζουμε για τις δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65-21 ο εισηγητής για την κοινωνική συνοχή, την προώθησή της απέναντι σε δεινές καταστάσεις στόχιας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 καταπίπτει αυτή 65-15 του εισηγητή πιλωτικό πρόγραμμα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ατομικό επίπεδο υπέρ κατά αποχές για να αλλάξουμε ηλεκτρονικά 6515 15 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίες. 22 υπέρ, 14 κατά, η αποχή μία εγκρίνεται. 65-43 καταπίπτει, 65-22 για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 65-23 εισηγητή το Ίδρυμα για την Εκπαίδευση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε 65 του εισηγητή για το αποθυματικό ακριβώς αυτό το ταμείο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι ολοκληρώσαμε με τους αριθμούς μας που πάμε τώρα στην νομοδότηση, παράγραφος 1, τροπολογία 1 του Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, παράγραφος 1, τροπολογία 2 του ιδίου, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, παράγραφος 2, τροπολογία 3 του ιδίου, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, παράγραφος 3, τροπολογία 4, Σαριασαγέ, εισηγητής κατά, υπέρ, κατά αποχές ε, εγπορύπτεται 5 δαρδέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραφος 6. Δύο οι ε, για διαγραφή. Εδώ όμω καταπίπτουν αυτέ γιατί την 65-16 την εγκρίνουμε λοιπόν καταπίπτουν οι άλλε. Παράφο 7, 8 Νταρντέν υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 9 του ιδίου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 10 του ιδίου, σε δύο μέρη, ξεχωριστά, χωρίς το ευαίσθητο ευάλωτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και για το ευάλωτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10, 12 τροπολογία μεγαλύτερη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ο 11 Φιλιππινιούν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα μισό λεπτό μισό λεπτό η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν θέλετε ναι αλλά όχι να στραφούμε και κατά της πλειοψηφίας Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοδότησης. Παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν. Συγητή και αναπληρώτρια Και τώρα ψηφορία για τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προπολογισμού για την κοιτοποίηση ακριβώ αυτού του ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση από τη στιγμή που πρόκειται για ιταλικό θέμα εδώ για την τετομάζω την αυτοκίνητο βιομηχανία αυτή τη γνωστή την ιταλική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάλι Ιταλική περίπτωση αλλά είναι για την περιοχή της Λομβαρδίας, στη Βορειοιταλία υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τι άλλο έχουμε. Όχι. Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτομία ο τίτλος δεν είναι σωστός όμως. Είναι η συμφωνία στο τελικό επίπεδο με το Συμβούλιο για την έκθεση που θα ψή αλλά easy αυτός είναι ο νέος τίτλος η Γίτα Στράινρουκ ήταν η συγγητριά μας γι' αυτό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για τη συμφωνία στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων Ιουλίου που μας πέρασε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και αν ψήφισαν όλοι, τότε πέρασε τις ψηφοφορίες. 34 υπέρ, 2 κατά, η αποχή μία. Και πάλι συγχαρτήρια στην εισηγήτριά μας και στους υπόλοιπους που προχώρησαν στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και ποια ήταν τα μέλη, δεν βλέπουμε εδώ. Πάμε τώρα στο σημείο 9. Τι πρέπει να ψηφίσουμε. Το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Όμεν Ρόιτεν για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρόκειται για τη βελτίωση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου με κανόνες δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται στην απασχόληση. Στην Νομική Επιτροπή με το κείμενο αυτό η Εύρυν Ρέγνερ είναι η, η Εβελίνα Ρέγνερ, ναι, είναι η συγκήτρια. Παράγραφος 1. Μισό λεπτό. Η συγκήτρια έχει το λόγο. Hetzelfde willen. Dat is de positie van de werknemerspartij om die te versterken. Dat is één. Επιθυμούμε να ενισχυθεί η θέση των ε, εργαζομένων και οι δύο μας, αλλά δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την παράγραφο 4. Για μένα η παράγραφος 4 είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατέβαλα μία προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τα όσα επιθυμεί η κυρία Ρέκνερ και υπάρχει και η τροπολογία 6. Την υποστηρίζω. Θα ήθελα να ζητήσω από τη σοσιαλιστική ομάδα τώρα να απόσχει στην ψήψη της παραγράφου 4. Τα δύο τρίτα των τροπολογιών της κυρίας Ρέγνερ τις δέχτηκα. Τα δύο τρίτα θα πρέπει κάτι να προσφέρει και εκείνη σε αντάλλαγμα. Κυρία Πρόεδρε, αυτό υποστηρίζω. Και με κοιτάζουν και με ρωτάνε τι σημαίνει η παραφός 4. Ποια είναι η διαφορά απόψεων ανάμεσα στην κυρία Ρέγνερ και σε μένα. Όταν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Υπάρχει πάντα το θέμα το τόπος απασχόλησης ενός εργαζομένου και χρειάζεται μια σχετική διαδικασία όχι στην Ολλανδία και όχι με την εφαρμογή του Ολλανδικού δικαίου. Κανένα απόψή μου δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι και υπέρ του εργαζόμενου. Και εγώ μίλησα και με γνώστες του θέματος. Θα πρέπει να είναι αρμόδιο το δικαστήριο εκεί που είναι η έδρα της εργασίας και όχι του εργαζομένου. Διαφορετικά θα ήταν κάπως παράξενη η νομική κατάσταση όπως θα εμφανιζόταν. Καλώς. Σημειώνω ότι με εισηγήτρια την κυρία Μενρόιτερ και συζήτηση πριν από την ψηφοφορία σε μια κατάσταση άκρος έκτακτη αλλά δεδομένου ότι κατάσταση είναι ακριβώ έκτακτη. Θα πρέπει να δώσω το λόγο και στο συντονιστή των σοσιαλιστών που μου τον ζητάει. Η κυρία Ρόιτερ, Ρόιτεν ε, κάνει λόγο για τις θέσεις της κυρίας Ρέγνερ, αλλά δεν είναι εδώ η κυρία Ρέγνερ για να απαντήσει. Νομίζω ότι όλοι έχετε στα χέρια σας τα έγγραφα που έχουν διανεμηθεί. Πρόκειται για τροπολογία υπαριθμών 9 στην νομοδότηση που αφορά την τέταρτη παράγραφο η εισηγήτρια προτείνει με το κείμενό της να χορηγηθεί αρμοδιότητα, δυνατότητα στον εργαζόμενο να ε, οχλήσει τον εργοδότη στο κράτος της απασχόλησης, ενώ η κυρία Ράιγνερ μιλάει για το κράτος της διαμονής του εργαζομένου. Άλλες παρεμβάσεις υπάρχουν, άλλες τοποθετήσεις. Όχι, θα ακούσουμε το μόνο τον κύριο Σέρκας για να συνεχίσουμε μετά. Η τελική ψήφος των σοσιαλιστών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απάντηση κυρία Σόιμεν Ρόιτε για την τροπολογία 9, αλλά και την 6, την 7 και την 8. Πρόκειται για αιτήματα λογικά ο εργαζόμενος να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στην, σε, έναντι μιας επιχείρησης στη χώρα στην οποία διανεμένει. Ε, σε χιλιάδες ε, περιπτώσεις ε, απαιτείται από τους εργαζόμενους όταν έχουν αποσπαστεί, όταν έχουν μετακινηθεί να επιστρέψουν στην αρχική τους χώρα για να ε, προσφύγουν στην δικαιοσύνη, για να προασπίζουν τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που ζητάμε. Ε, οι 6, 7 και 8 όμως είναι εξίσου σημαντικές για τις εργασιακές σχέσεις και είναι απόλυτα λογικές και μετριοπαθείς. Αν δεν γίνουν δεκτές θα ψηφίσουμε κατά στην τελική ψηφοφορία. Κύριε δεν μπορεί να ξανανοίξει τώρα συζήτηση. Μα κυρία Πρόεδρε, σε μια προσπάθεια να προτείνω λύσεις και να υποχωρήσω κάποια θέματα για να προχωρήσουμε. Τις τροπολογίες 6 και 8 τις υποστηρίζουμε. Είναι καλές τροπολογίες. Για την 9 δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε διότι οι εμπειρογνώμονες με τους οποίους, τον οποίο έχω στήσει τη γνώμη και οι εκπρόσωποι των διασυνοριακών εργαζομένων ε, θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί διαφορετική λύση. Τροπολογία νέα, λοιπόν. Το μικρόφωνο της ομιλήτριας δεν είναι αναμένο. Δεν είναι αναμένο το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Δεν ακούμε την πρόεδρο. Δεν ακούγεται η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Τροπολογία ένα Ρέγνερ. Και ράπτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνατε. Μετά την παράγραφο α. Τροπολογία 2 των αυτών συντακτριών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Μετά την παράγραφο α, ένα μάλλον, της κυρίας Στάινμπρουκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος πρώτη, τέσσερα, Ρέγνερ και Ράπτη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι, των αυτών συγκεκριών υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία Τροπολογία Επτά των δύο κυριών και της κυρίας υπέρ. Προκυπέρ. Κάτα. Άποχες. Απερίφθη. Τρίτη παραγραφός. 8η τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτη Ένα τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε την εννέα. Tout Ψήφισαν όλοι πέρα στις προφορίες. 19 υπέρ. 17 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται. Το σύνολο της νομοδότησης ηλεκτρονικά παρακαλώ. Υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία λέει η πρόεδρος. Ψήφισαν όλοι πέρας. Τριάντα υπέρ δύο κατά τέσσερις εποχές και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελειώσαμε λοιπόν αυτές τις ψηφοφορίες και κερδίσαμε και λίγο χρόνο. Μπορούμε όμως να περάσουμε στο σημείο 10. Δίνω το λόγο στην κυρία Edith Power. Α, όχι. Όχι, όχι, αλλά έχουμε αλλάξει τη σειρά. Σημείο 12. Όπως είχαμε πει και πιο πριν. Η κυρία Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ για να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμόνιες υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδές ανταλλαγές μαθητών, την έμισθη ή άμισθη κατάρτιση, την εθελοντική εργασία και την απασχόληση ως εσωτερική άμιστη βοηθή παρένθεση ΟΠΕΡ. Πρόκειται για σχέδιο οδηγίας, αναδιατύπωση συγκεκριμένα, της οδηγίας για την οποία προτείνει 77 τροπολογίες η εισηγήτρια, στην οποία και δίνω το λόγο, παρακαλώ. Μάλλον, ε, παρακαλώ οι συζητήσεις, παρακαλώ, παρακαλώ οι συζητήσεις να σταματήσουν. Οι κατηδίαν συζητήσεις να πάψουν, παρακαλώ. Κύριε Παπαδοπούλου, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τους γενικούς ε, στόχους της τρέχουσας πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανταποκρίνεται στην εντολή της δίνοντας ένα επιπλέον εργαλείο για την ενίσχυση κοινωνικής πολιτιστικής ε, ανταλλαγής και επαφών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, παίρνει τη μορφή οδηγίας που αναδιατυπώνει και τροποποιεί την οδηγία, τις οδηγίες ε, οι οποίες είχαν τα ίδια θέματα και καλύπτει έτσι τις ελλείψεις και τα προβλήματα ανάλογα και με την ε, λογοδοσία που έχει παρακολουθήσει και τις εκθέσεις που έχουν παρακολουθήσει αυτές τις εκθέσεις. Έχουμε λοιπόν ε, με δεδομένες τις προκλήσεις δημογραφικής αλλά και οικονομικής φύσεως που γνωρίζουμε την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσελκύσει υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό, νέους ε, από τρίτες χώρες και να διευκολύνει την ε, διακίνηση ε, διανιών από και προς τρίτες χώρες. Ερευνητές λοιπόν, φοιτητές, μαθητές, μη αμοιβόμενοι ασκούμενοι είναι οι κατηγορίες οι οποίες συμπληρώνονται με άλλες δύο κατηγορίες, τους αμοιβόμενους ασκουμένους και τις ε, μη αμοιβόμενες εσωτερικές άμυστες, ε, τις εσωτερικές άμυστες βοηθούς, τις ΟΠΕΡ όπως ονομάζονται. Όπου όμως δεν υπάρχει σαφής ορισμός και δεδομένου Δεδομένη τη απουσία αυτή ενό αφού νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να υπάρξει, ε, να προκύψει ο πειρασμό για την υπερβολική εκμετάλλευση αυτών των αμύστων εργαζομένων και ε, βοηθών. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι επιπλέον των πολύ στενών χρονικών περιοθωρίων για την κατάθεση αυτής της εκθέσεως ε, μέσα στα, στις διακοπές ε, του θέρους, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη μεγάλη πρόκληση, ότι δηλαδή ούτε είναι συγκεκριμένο, ούτε είναι επακριβές το πλαίσιο και δεν προσφέρεται ένα πλαίσιο ακριβές και συνεκτικό το οποίο να ε, προσδιορίζει τους όρους με τους οποίους θα έρχονται οι υπήκοοι τρίτων κρατών να ε, εργαστούν, να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι και περισσότερες ε, διαφορές εντοπίζονται ως προς την αντιμετώπιση των υπηκών τρίτων κρατών και δεν εντοπίζονται τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Διερωτώμεθα λοιπόν, οι ερευνητές, οι ΟΠΕΡ, οι ασκούμενοι μπορούν να βγουν από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και να ενσωματωθούν, θα ζητήσουμε αυτό δηλαδή στην Επιτροπή, σε μια νέα οδηγία. Ή αλλιώς θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε έτσι το κείμενο ώστε να συμπεριλάβουμε στοιχεία που θα καλύπτουν όλα τα, όλα τα κενά ε, και θα, θα επιτρέπουν ένα επαρκές επίπεδο εναρμόνισης ανάλογα με αυτό που απαιτείται στις οδηγίες όπως με την ενιαία άδεια Blue Card ή με τις συζητήσει που αφορούν τους εποχιακούς εργαζομένους. Αυτές ήταν οι δύο μας επιλογές. Επιλέξαμε τη δεύτερη λύση, αντιλαμβανόμενη βεβαίως πλήρως ότι είναι αναγκαία η απλούστευση και ο προσδορισμός αδρών γραμμών λύσεων και επιλογών στον τομέα αυτών, θεωρώντας όμως ταυτόχρονα ότι με δεδομένη την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια κοιτώντας την πλευρά του εργαζομένου περισσότερο, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας φάνηκε πολύ ε, ασαφές. Και γι' αυτό Δεδομένου ότι βλέπουμε ότι αναμειγνύονται διάφοροι τύποι απασχόλησης, διάφορες συμβάσεις απασχόλησης, ε, τύποι ερευνητών κτλ ε, και εργαζομένων δεν μπορεί να ενισχύσει τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων και την κοινωνική προστασία. Γι' αυτό ε, καταθέτουμε 77 τροπολογίες με αρκετές αλλαγέ οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν την πρόταση και να ενισχύσουν τους στόχους της και να υποστηρίξουν τους στόχους της. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε τις αγορές εργασίας για, καλύτερη, ε, για προσέλκυση καλύτερων δεξιοτήτων ανάλογα με τι ανάγκε τη αγορά. Δεύτερον, θέλουμε να αποφύγουμε κάθε είδου διάκριση ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Τρίτον, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα επαρκέ επίπεδο κοινωνική προστασία και ιδιαίτερα για την κατηγορία των ομπέρ. Και επίση, θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την κατηγορία της εξειδικευμένης, ε, του εξειδικευμένου εργαζομένου και επιπλέον θέλουμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στα μέλη της οικογενείας των ε, θέλουμε σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβαση στα μέλη της οικογενείας των εν λόγω εργαζομένων να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας. Δεν μπορεί αυτή να παραγνωρίζεται. Δεν είμαστε πεπισμένοι δε ότι οι ευρύτατες ε, διατάξεις οι οποίες ε, ισχύουν στο παρελθόν πρέπει να είναι υποχρεωτικές δεδομένου ότι η κοινωνική και δημογραφική κρίση έχει αυξήσει σημαντικά το χάσμα μεταξύ ε, Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών. Μεγάλες αποκλήσεις εμφανίζονται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, Ήπειρο και γι' αυτό το λόγο ζητούμε να ε, γίνει σεβαστή επαρκώς η αρχή της επικουρικότητας. Έχουμε καταθέσει 77 τροπολογίες και καλώς ορίζουμε ή αδίποτε άλλη τροπολογία. 20 Σεπτεμβρίου είναι η αδιποτε αλλη τροπολογια 20 σεπτεμβριου ειναι η για την κατάθεση τροπολογιών. Γίνεται συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές ε, για να δούμε τις θέσεις τους και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, Σαγιά. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η πρόταση Κομισιόν ε, γενικά είναι θετική. Χρειαζόμαστε περισσότερου καταρτισμένους ανθρώπου. Ε, βελτίωση των συνθήκων μετανάστευση είναι επίση καλό ε, στόχο και βοηθάει και τι αναπτυσσόμενες χώρε μακροπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά του ε, φοιτητέ και του μαθητέ δεν βλέπω σημαντικά προβλήματα. Η πρόταση ακολουθεί τι ισχύουσε οδηγίε έτσι κι αλλιώ παίρνουν συνήθω άδεια εργασία οι προτάσεις είναι, επίσης είναι πολύ σημαντικό εκεί που υπάρχουν ακόμη πιο θετικές διατάξεις να μπορούν να διατηρηθούν. Θα πρότεινα να διαγραφεί λοιπόν το τελευταίο τμήμα του άρθρου 4.2. Είναι σημαντικό η οδηγία αυτή να μην πλήττει τις χώρες οι οποίες έχουν πιο θετικές ε, διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των των φοιτητών δεν θα πρέπει να είναι πολύ περιοριστικό. Η σχέση αυτή τη οδηγίας με άλλα νομοθετικά κείμενα ε, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί. Υπάρχουν προβλήματα ενδεχομένω αν υποτεθεί ότι υπάρχει ε, όταν, όταν προϋποθέτει υποτίθεται ότι υπάρχει ε, σχέση εργασίας ε, ανάμεσα στο Ίδρυμα και τον ε, φοιτητή. Ε, μέχρι τώρα ε, οι, τα κράτη-μέλη μπορούσαν να περιορίσουν τα, τις κοινωνικές παροχές μόνο στις, αν να τις περιορίσουν έτσι ώστε να ισχύουν μόνο όταν υπάρχει σύμβαση εργασίας. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ε, το, τα ερευνητικά κέντρα σε, μέχρι σε ποιο βαθμό είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές παροχές αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας αυτή τη στιγμή. Το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο από την πρώτη μέρα εργασίας, ε, από την πρώτη μέρα άφηξης για να παρέχεται για παράδειγμα στέγαση ή το... Ε, το ερευνητικό κέντρο είναι υπεύθυνο για ασφάλιση εναντί ατυχημάτων αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασία. Αν δεν είναι αυτό υπεύθυνο, ποιο είναι υπεύθυνο. Δεδομένου ότι αυξάνονται οι δυνατότητε μετακίνηση, ε, θα πρέπει οι διαδικασίε να μην, να μην γίνουν υπερβολικά περιπλοκές. Πώ θα επηρεάσει η πρόταση την εγγύηση νεότητα, Πώς θα ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ή ε, ε, το, ε, οι σπουδέ κοστίζουν πολύ ενώ σε άλλες είναι δωρεάν. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για τη, από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι μια χώρα με υψηλές κοινωνικές παροχές που βασίζονται στη μόνιμη διαμονή. το βασικό πρόβλημα είναι οι προτινόμενες καινούργιες κατηγορίες ε, θελοντές, οπέρ κλπ. και το γεγονό ότι θεωρούνται ε, συμβάσει εργασία. Αν θεωρηθούν συμβάσει εργασία από, στην νομοθεσία μας δημιουργείται μια μεγάλη γκρίζα ζώνη. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ε, ίσως ε, θα καταλήξουμε σε εργατικό ντάμπινγκ και κάποιοι θα εκμεταλλευτούν υπέρ τους αυτές τις διατάξεις. Ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τις ΟΠΕΡ βλέπω. Ακόμα και αν συμπεριληφθούν οι ΟΠΕΡ, πιστεύω ότι ο βασικός σκοπός της οδηγίας δεν είναι να καλύψει τις ΟΠΕΡ. Για παράδειγμα, ε, θέλει η συγκεκριμένη να υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών προκειμένου να προσληφθεί ο ΟΠΕΡ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τόσο λεπτομερή νομοθέτηση για τέτοιου είδους ζητήματα. Ε, θα προσπαθήσω να συνεργαστώ πολύ θετικά με την ε, συγγήτρια και με τους άλλους και συγγητέ. Είναι σημαντικό αυτές οι καινούριες κατηγορίες να μην τύχουν εκμετάλλευσης. Ε, Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να εξαφανίσουμε την καλύτερη αντιπροστασία προστασία αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Μπενάρα Μπατού. Euh, Το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, συνδέεται με την πολιτική γειτονία. Ε, θέλουμε να την ανανεώσουμε, ιδιαίτερα με τις χώρες της ε, νότια Μεσογείου. Την περιμένουν πολύ. Είναι μια έκθεση που μας επιτρέπει να βγούμε από την παλιά νοοτροπία ότι οι μετανάστευς θα μας βυθίσουν. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο κινητικότητας. Αυτή είναι η καινούργια νοοτροπία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους, τη μαθητεία και τη ΟΠΕΡ, καθώ επίση και τους εθελοντέ, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νομικό πλαίσιο. Ειδικά για τις ΟΠΕΡ, για παράδειγμα, ε, αφορά κυρίω κοπέλες και είναι σημαντικό να επιτρέψουμε σε περισσότερες κοπέλες να έρθουν και να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Η Εύα Τζόλι, για παράδειγμα, συνάδελφός μας, ήρθε στη Γαλλία ως οπέρ για πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική εμπειρία για πολλά κορίτσια, για πολλές γυναίκες. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε νομικό πλαίσιο που να καλύπτει ε, αυτή την ε, μετακίνηση. Να επιμείνω στο εξής. Είμαι μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ε, ε, υπάρχει ένας αριθμός προγραμμάτων, τέμπους, έρασμους, μούντους κλπ. Που, μέσω των οποίων τα κράτη-μέλη δεν είναι συνεπή. Ε, ε, έχουμε εταίρους που ήταν σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Tempus και οι συμμετέχοντες ε, από πανεπιστήμια τουρκικά για παράδειγμα δεν κατάφεραν να έρθουν στην Ευρώπη ε, γιατί δεν τους δίνεται θεώρηση. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, να ακολουθούμε ένα νέο σύστημα με τις θεωρήσεις. Από τη στιγμή που κάποιος ε, συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ε, πρέπει να έχει δικαίωμα αυτομάτως να πάρει βίζα. Για να έρθει να συνενθεί με τους εταίρους κλπ. Όπως ακριβώς κάνουν και οι Ευρωπαίοι, όπως ακριβώς και οι Ευρωπαίοι εταίροι πηγαίνουν στη χώρα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. όταν κάποιο ε, συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει αυτομάτως να παίρνει βίζα. Μήπως κάποιος επιθυμεί το λόγο παρακαλώ. Όχι, κανείς. Ίσως η Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι συγγητές υπογραμμίζουν, πιστεύω, ότι υπάρχουν ε, τομείς που υποστηρίζουν την πρόταση, όπου μπορούν να υποστηρίζουν την πρόταση, όταν πρέπει να υπογραμμίσουμε το γιατί χρειάζεται αυτή η πρόταση. Έχουμε κάνει εκθέσεις υλοποίηση των σχετικών οδηγιών για τους φοιτητές. Έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις οδηγίες και η αναδιατύπωση που προτείνουμε στόχο έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Και έτσι από τα συμπεράσματα των ομάδων που έχουν καλύψει τις προτάσεις αυτές βελτιώνουμε και την ελκυστικότητα για ομάδες υπηκών τρίτων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις ομάδες τώρα, φοιτητέ και ερευνητές που ήδη προβλέπονται, δεν βλέπω να αμφισβητούνται πολλά από τις προτάσεις. Για τις νέες ομάδες πάντως, ιδιαίτερα για τους αμοιβόμενους ασκουμένους και τις άμυστες οικιακές βοηθούς επισημαίνεται κάποια προβλήματα, χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις, κυρίως σε στοιχεία που απαιτούν συμπληρωματικέ προποθέσει για την αποδοχή των αμύστων οικιακών βοηθών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνιση. Πάντως διατηρούμε μια, ένα ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με τις προτάσεις και των κρατών μέλων στο Συμβούλιο στι πραγματεύσει, για να επεκταθεί ο κατάλογος των προποθέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται και εφόσον αυτό ζητήσει και ο συνομοθέτης για τους αμοιβωμένους, για τους εμείς τους ασκουμένους και τις λοιπές κατηγορίες ε, δεν προτείνεται εναρμόνιση για το αν θα θεωρούνται εργαζόμενοι ή όχι. Σωστά το επισημαίνεται. Και αυτό γιατί η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν η εναρμόνιση. Αλλά το να επαφεθεί στο κάθε κράτος μέλος η απόφαση του εάν ο έμισθος ασκούμενος λογίζεται ως εργαζόμενος ή ως φοιτητής ή ασκούμενος εφόσον προβλέπεται ένα τέτοιο καθεστώς στη νομοθεσία του, του κάθε κράτους μέλους. Για την κινητικότητα, διατάξεις είναι πολύ σημαντικές. Θα έχετε ασφαλώς υπόψη πώς συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, ιδιαίτερα για τις μετατάξεις ε, και αποσπάσεις εντός της ίδιας επιχειρήσεως του ίδιου και αντίστοιχα θα δούμε τι είδους προτάσεις μπορούν να προκύψουν και να αξιοποιηθούν και στις δικές μας, στη δική μας περίπτωση, στις ομάδες αυτές δηλαδή της οδηγίας. Ένα άλλο θέμα που επισημάνθηκε πολύ σημαντικό είναι η σχέση της οδηγίας με την ενιαία άδεια. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Blue Card, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να παραμείνει το Single Permit ε, όπως έχει και εξαιρέσει να προβληθούν μόνο όπου και μόνο απαιτείται. Αυτή είναι η προσέγγιση της Επιτροπής. Ως προς την πρόσβαση στην αναζήτηση θέσεων εργασία, για φοιτητέ, πτυχιούχους, για ερευνητέ που έχουν κλείσει ένα κύκλο ερευνητικό, θα ήθελα να υπογραμμίζω ότι πρόκειται για πρόσβαση στην αναζήτηση θέσεων εργασία και όχι πρόσβαση στην αγορά εργασία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το ε, εν λόγω κράτο μέλος ε, το οικείο κράτο μέλο δώσει τη σχετική άδεια. Δεν δίδεται δηλαδή αυτομάτω άδεια πρόσβαση στην αγορά σε κάποιον που έχει ολοκληρώσει τι σπουδέ του ή που έχει κλείσει ένα ερευνητικό κύκλο. Και ξέρουμε βεβαίω πόσο σημαντικέ προκλήσει και δυσκολίε αντιμετωπίζουν λόγω τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κάποια κράτη-μέλη. Αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Μια τελευταία λέξη. Το άρθρο 79.5 της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζει τους όγκους υποδοχής υπηκών τρίτων κρατών δεν παραβιάζεται γιατί εκεί ορίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι εκείνες οι οποίες θα δώσουν την, θα λάβουν την απόφαση για το πόσοι πει ή τρίτων κρατών μπορούν να γίνουν δεκτοί. Δεν αλλάζουμε λοιπόν τους αριθμούς των υπηκών τρίτων κρατών που θα υποδεχθεί ένα κράτος μέλος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ την εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, για, ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Να κάνω και εγώ μερικά σχόλια. για τις ε, προτάσεις του ΕΛΚ. Ναι, περιμένουμε και εμείς ε, να ε, το συζητήσουμε. Μερικά από τα σχόλια σας μας με βρίσκουν σύμφωνοι. Ο ορισμός του φοιτητή δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα νομίζω. Τα βασικά προβλήματα αφορούν τις δύο καινούριες κατηγορίες. Τους έμιστους φοιτητές και τις ΟΠΕΡ. Ε, τους έμιστους μαθη... υπομαθητεία και ε, τους, ε, τις ΟΠΕΡ. Εκεί θα κάνουμε τις τροπολογίες μας, θα τις εστιάσουμε. Είπατε ότι στο άρθρο 21.1 ε, ε, ορισμένοι περιορισμοί ε, θα πρέπει να ξαναειδωθούν, να ξανακοιταχτούν. Εδώ έχουμε διαφορετικές γνώμες μεταξύ των κρατών μελών. Δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια προσέγγιση. Και στο Συμβούλιο πιστεύω θα συζητηθεί πολύ το θέμα γιατί ό,τι είναι καλό για, το, ε, για τους ε, Σουηδούς, ε, για το σουηδικό μοντέλο, δεν είναι εξίσου καλό ενδεχομένως στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού. είναι δευτερεύοντα θέματα, θα πρέπει να συζητηθούν πολύ. Ε, συγγνώμη, δεν είναι δευτερεύοντα θέματα και θα πρέπει να συζητηθούν πολύ. Τώρα, ποιο είναι υπεύθυνο ε, στι περιπτώσει κινητικότητα και πώ θα επηρεαστεί η πρωτοβουλία νεότητα, η εγγύηση νεότητα, είναι και αυτά δικά, είναι και δικά μου ερωτήματα. Ε, σίγουρα θα πρέπει να αποφευθεί το dumping. Ε, σε ό,τι δεν αφορά την οικογενειακή ε, πανένωση δεν ήθελα να επισέλθω στο θέμα. Αυτό είναι θέμα τεχνοκρατών. Αλλά αν η Κομισιόν μας υποβάλλει πρόταση που θα αναδιατυπωθεί και επειδή είναι αναδιατύπωση θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ περιορισμένη <laughs> έχουμε όμως τεράστιες αλλαγές και χωρίς ε, κοινό κανονισμό και κοινή νομική βάση για όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να δούμε πώς θα κλείσουμε τα κενά. Οπότε περιμένω και εγώ να συζητήσουμε μαζί σας. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες κύριε Σατού. Ε, γνωρίζω ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Στόχος είναι να διευκολύνει την ελευθερία μετακινήσεων, κυκλοφορίας, γιατί κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και τους ε, πολίτες τρίτων χωρών και τους πολίτες Ευρώπης, και πολιτιστικές ανταλλαγές κλπ. Δεν συμφωνώ με το θέμα της τουρκικής θεώρησης, των τουρκικών θεωρήσεων. Είναι πολύ πολιτικό θέμα. Συζητείται στην κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή, στη μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή. Είμαι μέλος αυτής της επιτροπής και λειτουργεί ε, ε, προς τις δύο κατευθύνσεις. Και η Τουρκία θα πρέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε πολλά θέματα, αν θέλουν να πάρουν αυτά που ζητούν για την βίζα. Αυτό είναι πολύ πολιτικό θέμα. Το θέμα συζητείται ε, στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή πολύ. Τέλος, ελεύθερη κυκλοφορία η ελεύθερη κυκλοφορία είναι το υπαριθμόν ε, ε, ένα στοιχείο της, ε, του κοινωτικού κεκτημένου. Θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και εγώ ως μετανάστης από την Κύπρο ε, ξέρετε ότι ε, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Τουρκία δεν μου επιτρέπει να πάω στο, ε, σε ένα κομμάτι της χώρας μου. Μου αρνείται λοιπόν το βασικό μου αυτό δικαίωμα. Συνεπώς, αν θέλουν ελευθερία κυκλοφορίας θα πρέπει οι Τούρκοι να σέβονται και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και να σταματήσει να τα παραβιάζει στη χώρα μου. Το θέμα αυτό όμως δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας. Ε, ε, είμαστε η γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι Δημοσίων Ελευθεριών, που είναι εκείνη επί της αρμόδια. Για τις τροπολογίες η προθεσμία, έχουμε στα αγγλικά μόνο μάλλον τις τροπολογίες, και με ηλεκτρονικές υπογραφές, ψηφιακές αν θέλετε. Όχι ηλεκτρονικές, ψηφιακές, έτσι, διαφορά ανάμεσα στα δύο. 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12 και 18 μετά 28, 25 την βαστική ε, λύση 26 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και 17 Οκτωβρίου Επιτροπή. Δημοσίων Ελευθεριών και μετά πάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 10 με την Edith Bauer που θα λάβει το λόγο και η οποία θα μας παρουσιάσει το της για τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων παρέχοντας τους εργαζομένους ε, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών. Οι Επιτροπές Γυναικών και Αναφορών Αυτές οι δύο επιτροπές θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Κύριε Μπάουερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι ο λόγος για την γενετικότητα. Αλλά αποκλειστικά πλέον για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαίρουν της, του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάσταση για απασχό για εργασία σε τρίτες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μόνο 3,1% των εργαζομένων, από ό,τι μας λένε οι στατιστικές του 2011, ε, αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή που τους προσφέρεται. Το Ευρωμαρόμετρο δείχνει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επισημαίνουν πολύ μεγάλο αριθμό εμποδίων στη διακίνηση και εργασία σε άλλο κράτος. Υπάρχει βέβαια ο κανονισμός 492, ο οποίος ισχύει. Η εν λόγω οδηγία ενισχύει τον κανονισμό. Αυτός είναι ο στόχος της. Το κύριο ζήτημα βέβαια είναι γιατί να χρειαζόμαστε την ενίσχυση του κανονισμού όταν θεωρητικά έπρεπε να εφαρμόζεται απευθείας και αμέσως. Η ευρύτερη απάντηση νομίζω είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για το πώς μπορούν να ενισχυθούν ε, κάποια σημεία επικοινωνίας, επαφής, ενημέρωσης, υποστήριξη εκείνων που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλη χώρα και που ενδεχομένως να δίνουν απαντήσεις σε προβλήματα. η οδηγία, ο κανονισμός μάλλον, ορίζει ποιες είναι, ποια είναι τα όρια της πρόσβασης αυτής, ε, τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνδικαλιστικά σωματεία, στέγη, ε, σχολεία για τα παιδιά, κοινωνικές συνθήκες και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι κάθε τροπολογία που θα γίνει δεκτή για την οδηγία δεν μπορεί να ξεπερνάει αυτό το ε, πλαίσιο που έχει οριστεί από τον κανονισμό. Εμείς προτείνουμε ένα πεδίο εφαρμογής που θα επεκτείνεται και στην αποκατάσταση στη θέση εργασίας η αποζημίωση για λόγους ανεργίας, τα όργανα των κρατών μελών οι σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως και στους υπηκόους και στους εργαζόμενους από άλλο κράτος μέλος. Και έχοντας ε, έρθει σε επαφή και ανταλλαγή απόψεων με το δίκτυο για την ισότητα ευκαιριών, θα ήθελα να επισημάνω ότι και αυτοί προσφέρουν δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες. Εθνικά λοιπόν σημεία επαφής και ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής θα πρέπει να συστήσουν τα κράτη-μέλη ώστε να καθίσταται πιο εφικτό το εγχείρημα της εγκατάστασης σε άλλο κράτος. Εάν, και αυτό μπορεί να συμβεί φαντάζομαι, αρμόδια, συναρμόδια είναι περισσότερα από ένα κράτη-μέλη, γιατί μπορεί να υπάρχουν ζητήματα υλοποίησης διατάξεων που επιμερίζονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ή επί παραδείγματι μπορεί να απευθυνθεί κάποιο σε μια υπηρεσία κράτου μέλου που δεν είναι όμω ε, ενήμερη ή εξοπλισμένη επαρκώς για να δώσει απαντήσει ε, στα αιτήματα για πληροφόρηση. Επομένω θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί και να συνεργαστεί με μια άλλη αντίστοιχη υπηρεσία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα της πολυγλωσίας και μέσα ε, και ενημέρωση για ένδικα μέσα και δυνατότητα αποκατάστασης ή διεκδίκησης ε, δικαιωμάτων. Και αυτό θα πρέπει να προσφέρεται και στους υπηκόους τρίτων κρατών, αλλά και στους οικείους υπηκόους, ενδεχομένως που θέλουν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος. Τεχνικές ε, προσαρμογές επίσης θα χρειαστούν. Το να χρησιμοποιείται δηλαδή η ίδια ορολογία και πάνω απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για μετανάστευση αλλά για κινητικότητα εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε επίσης να γίνει μια επαλήθευση με αντίστοιχες οδηγίες ε, που αφορούν ε, τα δικαιώματα των μέλων της οικογένειας, των ε, εργαζομένων σε κινητικότητα και λοιπά θέματα σχετικά. Και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω το ζήτημα της συλλογικής αγωγής, γιατί εδώ βεβαίως σύσταση είναι μόνο αυτό που διατυπώνω και δεν ε, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλά σε τις περιπτώσεις διεκδίκησης ε, δικαιωμάτων, άσκηση ξενδικών ε, μέσων, ε, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία η δυνατότητα για μια συλλογική αγωγή. Επίσης γίνεται μια παραπομπή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το άρθρο 45 Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πολλοί άριθμες είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που προσδιορίζουν τους ε, περιορισμούς του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετά καθαρή εικόνα για την ε, για τους λόγους που οδηγούν στην αδυναμία αυτή εφαρμογής του κανονισμού. Γι' αυτό και ζητούμε την κατάρτιση των ε, υπαλλήλων εκείνων, των ε, μελών των υπηρεσιών εκείνων του προσωπικού που καλούνται να υλοποιήσουν τον κανονισμό. Και όλα αυτά ολοκληρώνοντας ήθελα να πω ότι προσπαθώ πάντα να περιοριστώ στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας όπως είναι ορισμένο ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια για την παρουσίαση. Σε μεγάλο βαθμό ε, συμφωνώ. Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αποτελεί πυρήνα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και θεμέλιο λίθο της ε, ενωσής μας. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεν λειτουργεί πάντα όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αντιληπτό το πώς λειτουργούν οι κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων. Ποτέ δεν ήταν στόχος της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, να γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ε, εθνικότητες ή χώρες προέλευσης. Οπότε αυτή η πρόταση πρέπει να ειδωθεί ως ευκαιρία να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι δυνατότητες ε, οι εταιρείε να προσλαμβάνουν αλλοδαπό προσωπικό με δίκαιο τρόπο. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η πληροφόρηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι δεν ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματά τους. Ίσως σε πολλές χώρες τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους στη χώρα στην οποία θα μετακινηθούν. Γιατί πολλές φορές οι μετακινήσεις αυτές καταλήγουν σε κακές συνθήκες εργασίας για το εργατικό δυναμικό που μετακινείται. Στρεβλώνεται προφανώς και ο ανταγωνισμός με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολλή δουλειά εμείς και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι για το θέμα της ενημέρωσης. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν την πρωτοβουλία, να προασπίσουν τους εργαζόμενους που είναι μέλη τους. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν, όπως το άρθρο 4 Σε κάποια κράτη-μέλη τα συμβαλόμενα μέρη εγγυώνται ότι θα γίνουν σεβαστοί οι κανόνες και οι επαγγελματικές οργανώσεις δεν μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν την ειδική αυτή αναγνώριση. Η αναγνώριση αυτή δεν είναι σαφής ούτε στο άρθρο ε, ε, η ενημέρωση αυτή δεν είναι σαφή στο άρθρο 4 της Κομισιόν. Θα ήθελα να μας το εξηγήσει. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτή η αναγνώριση για να αποφύγουμε επίσης και αλληλεπικάλυψη των συστημάτων. Πάντως, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι η έκθεση είναι καλή και διευκρινίζει το κείμενο της Κομισιόν. Προσωπικά πιστεύω θα έπρεπε να πάμε λίγο πιο μακριά στο άρθρο 7 με τις ε, σελίδες στο ίντερνετ όπου εμφανίζονται πληροφορίες για τα δικαιώματα των αναζωμενών. θα πρέπει να διαθέτουμε ένα καλύτερο εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών κατά την άποψή μου. Ίσως ε, να εμβαθύνουμε, ε, να διευρύνουμε αυτά που ήδη έχουμε, αποφεύγοντας βέβαια την αλληλεπικάλυψη. Ε, σε γενικέ γραμμέ όμω συμφωνώ με την έκθεση. Σας ευχαριστώ, Μπενιόν. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε Κορνέλισεν, Becker πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μπάουερ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σίγουροι ότι ε, θα ε, καταργήσουμε τα βασικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή. Και το προσχέδιο έκθεσης έχει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και τροπολογίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε για παράδειγμα η συλλογική αποκατάσταση και οι βέλτιστες πρακτικές. Αυτό που ξεχάστηκε όμως είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα με σε περίοδο κρίσης, δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να διευρύνουμε το πεδίο μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους νέους για παράδειγμα, για να ασκήσουν και αυτοί τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, για παράδειγμα φοιτητέ, μαθητές. Γενικά όμως πιστεύω ότι είναι καλή έκθεση και θα συνεργαστώ με την συγγήτρια και τους ε, σκιώδης συγγητές. Κορνέλισεν και επόμενη. Um, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την καλή πρότασή της. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα μεγάλο κομμάτι της. Βέβαια και πάλι είναι λίγο ε, α, ε, απογοητευτικό που ε, δεν προσφέρει λύσεις εναντίον του στρεβλού ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης γιατί και πάλι ε, είναι νομικός ε, εφικτό να δίδονται χαμηλότεροι μισθοί στους ε, αποσπασμένους εργαζόμενους κλπ. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται να διευρυνθεί, να διευρύνεται επάπειρον, επαόριστον και επάπειρον το πεδίο. Τουλάχιστον κάτι γίνεται έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Η κυρία Μπάουρα έχει δίκιο που λέει ότι η έλλειψη πληροφόρηση είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια άσκηση των δικαιωμάτων. Οπότε η επαρκής κατάρτιση ε, των ε, δημοσίων υπαλλήλων ε, είναι μια καλή πρόταση. Όμως είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένοι και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να τους δίδεται πληροφόρηση σε μία γλώσσα που να καταλαβαίνουν, που να κατανοούν αυτό είναι σημαντικό να προσθεθεί. Ε, επίσης, οι φορείς που ασχολούνται με θέματα ισότητας έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διάκρισης, των διακρίσεων. Ε, θα πρέπει όμως να ε, έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα γι' αυτό. Θα ήθελα να προσθεθεί μια τροπολογία, θα υποβάλω μια τροπολογία αυτό το θέμα. Ε, ένα άλλο θέμα είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Ένα από τα εμπόδια στην άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων είναι ότι νομικό τα κράτη-μέλη ε, είναι υποχρεωμένα ε, να αναγνωρίζουν οικογενειακές σχέσεις που έχουν συναυθεί σε άλλες χώρες αλλά πολύ συχνά ε, δεν το κάνουν, για παράδειγμα με, ε, για τα παιδιά ή για ε, συζύγους, πρώην συζύγους κλπ. Ε, για την συλλογική αποκατάσταση είναι καλές οι προτάσεις Μπάουερ. Επίσης υπάρχει το δικαίωμα αν ένας εργαζόμενος κερδίσει τη δίκη να ε, αποζημιωθεί για ε, το εισόδημα το οποίο έχει απολέσει. Το απολεσθέν εισόδημά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλειβέτη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η στιγμή είναι κατάλληλη για μια παρόμοια ανάλυση με παρόμοιο θέμα και στο αν όλοι συμφωνούν ότι η ελεύθερη διακίνηση κυκλοφορία εργαζομένων ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ένωσή μας, πριν ε, από μερικές εβδομάδες ένα σημαντικός υπουργός εργασίας ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πορτοκαλί κώδικα ουσιαστικά στην αγορά εργασίας γιατί υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες που έρχονται κυρίως από τις ανατολικές χώρες. Ε, επικροτώ την άποψη της κ. Μπάβαρο θα πρέπει να, κάνουμε μια, να δούμε τη διαφορά μέσα στην μετανάστευση και στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Γιατί Υπάρχουν στιγμές κατά την άποψή μου που παρόμοια σχόλιο θίγουν ε, Ευρωπαίους πολίτες όπως τους Ρουμάνους στην περίπτωσή μας. Σημαντικό είναι λοιπόν να διαθέτουμε ένα νέο εργαλείο για τα δικαιώματα των εργαζομένων που κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος για την κινητικότητά τους ε, στις χώρες μας ε, και να κάνω μια ανάλυση κατάλληλη και να δούμε περισσότερο και καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα. Αυτός είναι και ο σκοπός μας άλλωστε. Η κυρία Λουμπέτσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 3% των ε, πολιτών που κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος ε, που μπορούν να μετακινηθούν και να δουλέψουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν έμπρακτα ότι αφορά μόνο λίγους εκλεκτούς παρόλο που κανονικά θα έπρεπε να αφορά όλους τους πολίτες. Και αυτό το δείχνει και η έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που λέει ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια για την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων. Επειδή ε, οι εθνικοί οργανισμοί δεν έχουν εντάξει ρυθμίσει Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κανονισμό τους και δεν είναι αρκετό αυτό και μόνο. Πρέπει κανείς να μπορεί και να το εφαρμόσει. Συμφωνώ όμως υποστηρίζει η κυρία Μπάουερ στην εκθεσή της για ορισμένα σημεία επαφής ε, και για ε, ε, ιστοσελίδες ε, που θα ενημερώνουν. Θα πρέπει να δείχνουμε, να ενημερώνουμε τους πολίτες που με τη σειρά τους θα λάβουν πληροφορίες για αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία τους και να τους λέμε ποια είναι, ποια είναι τα αρμόδια όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Πρόκειται για πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί επιτρέπουν οι πληροφορίες αυτές ε, στους πολίτες να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για τις δυνατότητές τους να μεταμούν στο εξωτερικό σε άλλες χώρες και να εργαστούν και οι πολίτες να διαθέτουν τη γνώση και να προετοιμαστούν καλύτερα πριν από την αναχώρησή τους ε, και να περιστούν και προβλήματα έτσι που θα αντιμετωπίσουν στην άλλη χώρα διοίκησης. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς και να προσέξει καλύτερα την ανάλυση αυτής της οδηγίας. Όλοι λένε οι εμπειρογνώμονες ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για να ξεφύγουμε από την κρίση. Αλλά την ευκαιρία αυτή θα πρέπει πραγματικά να την προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Κύριος Μπένιον, ευχαριστώ πολύ. λόγο. Πιστεύω πάντως ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μια από τις αρχές τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουμε και παρά τις δυσκολίες που μερικές φορές εντοπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών όπου λαϊκιστικές τοποθετήσεις του τύπου επηρεάζουν πολύ συχνά τους πολίτες μιας περιοχής, μιας χώρας ε, ότι, ε, και τους πείθουν ότι μπορεί να κινδυνεύει η δουλειά τους λόγω της ε, κινητικότητας κάποιων άλλων. Και αντί να αναζητήσουν οι ίδιοι λύσεις μέσα από τη δική τους κινητικότητα στην αγορά εργασίας, κατηγορούν όλους τους άλλους και όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να υποστηριχθεί η ιδέα και να υπογραμμιστεί η ιδέα ότι είναι υποφελής προς τους πάντες ε, το, η δυνατότητα της κινητικότητας και ότι δεν έχει μηδενικό αποτέλεσμα. Ε, δεν πρέπει να αφήσουμε να παρασύρονται οι πολίτες από το λαϊκισμό. Και πολύ σύντομα ένα σχόλιο. Ωστόσο, επί κυρία Κορνέλισσα, για τις οικογένειες, ότι υπάρχουν θέματα σε σχέση με τις χώρες Σέγγεν και μη Σέγγεν οι εργαζόμενοι οι οποίοι από τις χώρες εκτός Σέγγεν μεταβαίνουν σε χώρες Σέγγεν, εάν έχουν, ε, υπηκό, αν έχουν συζύγους υπηκόους ε, τρίτων κρατών, ε, αναγκαστικά εκείνοι θα πρέπει, εκείνες θα πρέπει να ζητούν θεώρηση διαβατηρίου τύπου Σέγγεν προκειμένου να μπορούν να ακολουθήσουν τους συζύγους τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ιδιαίτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και λόγω του, καθεστώ, του, του παρελθόντος της μεγάλης αυτοκρατορίας ε, πολύ πολλά είναι τα ζευγάρια τα μεικτά από τρίτες χώρες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα διότι ο, η, η σύζυγος τρίτης, υπηκός χώρας που θέλει να συνοδεύσει τον ή την σύζυγο ε, σε χώρα Σέγγεν υποχρεούται από χώρα μη Σέγγεν υποχρεούται να περνάει από τη διαδικασία της θεώρησης διαβατηρίου. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και το αντίστροφο, αλλά πρέπει πάντως να το κοιτάξουμε. Απλά και μόνο να υπενθυμίσω κάτι αποτελεί από τη σημαντικά κείμενα και ο Επίτροπος θα ήθελε να ολοκληρωθεί η πριν από τώρα σε ένα πλαίσιο που ο καθένας ε, έχει υπόψη του ότι το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων αποτελεί ένα από ε, τους ακρογωνίους λήθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τους πυλώνες ε, που θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω την εσωτερική αγορά. Παρακαλώ όμως προσέξτε όχι ότι όλη η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανεργία εδώ και εκεί στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα λυθεί το θέμα αυτό με την ε, κίνηση αυτών των εργαζομένων από την περιφέρεια προς το κέντρο είτε ότι δημογραφικά έτσι θα εξεταστεί και θα επιληθεί, επαναλαμβάνουμε το θέμα. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η ελεύθερη κυκλοφορία δηλαδή των εργαζομένων και τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και ανισορροπία ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια και με τον Υπουργό Υγείας της Λιθουανίας συνομίλησα χθες το βράδυ και ακόμα και στις περιφερειακές χώρες δημιουργείται ένα πρόβλημα ισορροπίας ανάμεσα στις διάφορες γενιές. Φεύγουν έξυπνα μυαλά και δεν μπορούν να αναπτυχθούν έτσι εύκολα οι περιφερικές χώρες με αυτούς που απομένουν. Είναι κόσμος ε, που έχει ξεκινήσει όμως από την άλλη μεριά να αναζητεί δουλειά στο κέντρο, εντάξει και αυτοί να έχουν δυνατότητες και ευκαιρίες, αυτό άλλωστε προτείνει το κείμενο του Επιτρόπου, αλλά το να θεωρεί κανείς ότι αυτή η μετακίνηση μακροοικονομικά θα επιφέρει μια ισορροπία στις οικονομίες ακριβώς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελούσε τρομερό λάθος. Καλό θα ήταν και εμείς να προσφέραμε, να βάζαμε ένα λιθαράκι στην οικοδόμηση αυτή, αλλά δεν είναι όμως μια λύση σε προβλήματα που διαφορετικά θα πρέπει να εξεταστούν γιατί αυτή την έκφραση εγώ χωρίς τα χρησιμοποιώ με διάθεση γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος, αυτό το θέμα της ελεύθερη πληροφορίας των εργαζομένων και άλλος ένας όμως όρος, έστω και αν δεν περιγράφεται στις συνθήκες, είναι το δικαίωμα του καθένα να παραμείνει στη χώρα του, να εργαστεί στη χώρα του και αφορά όσους ε, είναι στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα να έχουν και αυτό δικαίωμα εκεί να παραμείνουν να βρουν δουλειά. Εντάξει, πέρα τώρα από τον τεχνικό χαρακτήρα των σημερινών συζητήσεων, όλα αυτά μπαίνουν στα πλαίσια μιας γενικής πολιτικής που σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοούμε. Λίλιαν Μουρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά η εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Επιτροπή λοιπόν, Μουρ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Να απαντήσω εν συντομία στην ερώτηση κυρίας Μπάρακ. Γιατί είναι απαραίτητη η πρόταση Κομισιόν. Όπως όλοι σας αναφέρατε, η, ελευθερία των, η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων είναι θεμελιώδη αρχή του κοινωτικού νόμου. Ε, παρόλο ότι ισχύει και εφαρμόζεται εδώ και 40 χρόνια, η κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή. 3,1% ε, είναι η διαμεθουριακή διασυνοριακή κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη πρόταση. Ε, ένας λόγος είναι η διασυνοριακή κινητικότητα και η αύξησή της. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Οι υπηρεσίε της Κομισιόν λαμβάνουν μεγάλο αριθμό παραπώνων περί παραβίασης των δικαιωμάτων αζωμένων στην ελεύθερη κυκλοφορία. Με ελλειπή εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι οι εργοδότες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζόμενων και ακόμα πιο σημαντικό οι εργαζόμενοι ή αυτοί που αναζητούν εργασία δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζονται. Και οι, διάφορες, οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται με θέματα πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε ότι για παράδειγμα πέρσι ένας μόνο φορέας, η EuroAdvice, ε, έλαβε 10.000 αιτήματα πληροφόρησης για τέτοιου είδου θέματα. Οπότε πραγματικά ο στόχος της οδηγίας αυτής είναι, στόχος αυτής είναι να ε, δώσει ένα πλαίσιο καλύτερης πληροφόρησης και ενημέρωση. Με ένα φορέα ο οποίος θα βοηθάει σε κάθε χώρα τους ενδιαφερόμενους. Και όταν πρέπει να λυθεί μια, να, όταν πρέπει να προσβληθεί μια διοικητική απόφαση, όταν υπάρχει μια διαφορά, να βοηθάει. Ε, έγινε και μια ερώτηση, μάλλον μας ζητήθηκε να διευκρινιστεί το άρθρο 4 της πρότασης. Το άρθρο 4 της πρότασης εκφράζει ακριβώς αυτή την ιδέα, ότι δηλαδή αν ένας Εργαζόμενος κάποιος που αναζητά εργασία, έχει πρόβλημα και θέλει να προσβάλλει κάποια απόφαση ή να ε, φέρει μια υπόθεση στο δικαστήριο, θα πρέπει να τον συνδράμουν, να το συνδράμει κάποιος φορέας, κάποιο σύστημα. Συνεπώς χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα, ε, κάτι το οποίο μάλιστα είναι και μια ε, ρήτρα που εμφανίζεται και σε άλλα νομικά κείμενα που αφορούν θέματα ε, ισότητας, ε, οδηγία 2043 και στις ε, ε οδηγίες ε, φύλου, της ονομαζόμενης gender directives. Έγινε άλλο ένα σχόλιο για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ε, θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Η πρόταση αυτή καλύπτει και το άρθρο 45 της συνθήκης και τον κανονισμό, του 4, 492. Ε, καλύπτονται ό, οι, όσοι αναζητούν εργασία καλύπτονται από το άρθρο 45 της συνθήκης και ο κανονισμός 492 προβλέπει ίση μεταχείριση από τις εθνικές υπηρεσίες ε, προσφοράς εργασίας. Να σας κάνω και μερικά σύντομα σχόλια για τις ε, τροπολογίες που προτείνονται. Τροπολογία 1. Να επαναλάβω μια ανησυχία που, έχουμε, ε, που εκφράσαμε και νωρίτερα αυτή τη βδομάδα στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων Γυναικών. Η ε, τροπολογία 1 εισάγει τον Ε, τον ορισμό των μελών της οικογένειας κάνοντας αναφορά στην οδηγία 2004-38. Ε, αυτό όμως δημιουργεί τον κίνδυνο να μην καλυφθούν οι εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους. Γιατί, Γιατί η 2004-38 περιπικότητας δίνει το δικαίωμα σε έναν ε, πολίτη να μετακινηθεί και να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος. Όμως οι συγκεκριμένοι ζώμενοι μετακινούνται αλλά δεν ζουν σε μια άλλη χώρα, συνεπώς δεν καλύπτονται από τη 2438. Συνεπώς μας ανησυχεί το γεγονός ότι προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός του 2004, της Μπορεί να μην καλυφθούν με αυτόν τον ορισμό. Τώρα, τροπολογία 6. για, την, ε, ε, για τις ομαδικές ε, συλλογικές ε, ε, ε αποκαταστάσεις. το, η, έκθεση, η παράγραφος 15 του, της Ετωλικής έκθεσης αφορά την παράγραφο 4 ήθελα να σας πω. για την τροπολογία 11 η αλλαγή από migrant σε mobile, ε, ε, αντί για migrant worker να μιλούμε για mobile workers ε, στα αγγλικά. Ε, το έχουμε συζητήσει. η νομική μας όμως, η γλωσσομαθής νομική μας, μας είπαν ότι στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας και του άρθρου 45 συνθήκης η καλύτερη, ο καλύτερος όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η λέξη, είναι ο όρος migrant workers. Τροπολογία 12. που αλλάζει την τον όρο ελεύθερη κυκλοφορία σε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Στην παράγραφο 26 του, της έκθεση. Έκθεσης, η παράγραφο 26 συνδέεται με το άρθρο 8, παράγραφος 2. Το άρθρο 8, παράγραφος 2 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη όταν συστήσουν αυτά, αυτούς τους φορείς που θα βοηθούν τους ε, εργαζόμενους, ε, τους δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις αρμοδιότητες αυτού του φορέα έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και καθήκοντα γενικότερα υπέρ των, που να αφορούν γενικότερα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όχι μόνο εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο και μιλούμε για ελεύθερη κυκλοφορία και όχι μόνο ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Τελευταίο μου σχόλιο σχετίζεται με την τροπολογία 14 που αναφέρεται στο άρθρο 4 της πρότασης. Όπως είπα και προηγουμένως, η πρόταση Κομισιόν στο άρθρο 4 αναπαράγει μια ε, ε, ρήτρα η οποία ήδη χρησιμοποιείται ε, στις ε, οδηγίες για το φύλλο και στην οδηγία για την αποφύγη των διακρίσεων. Είναι στάνταρ. Ε, δεν μας πείθει έτσι κι αλλιώς η πρόταση ότι για το γεγονός ότι αλλάζει κάτι και ότι υπάρχει κάποιο όφελος που προκύπτει από το να αλλάξουμε αυτή τη ρήτρα η οποία είναι στάνταρ και εμφανίστηκε σε άλλα νομικά κείμενα. Ευχαριστώ. Εισηγήτρια. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Και τα σχόλια της Επιτροπής βεβαίως. Πολλά θέματα μπορούμε να εξετάσουμε και να αναλογιστούμε, αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε ότι αυτή η οδηγία αφορά ουσιαστικά την καταπολέμηση των διακρίσεων επί τη βάση της ηθαγένειας. Και ξέροντας ότι υπάρχουν και άλλοι, ε, άλλα νομοθετήματα, άλλες διατάξεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το δούμε επ' αυτή τη σκοπιά. Κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις συναδέλφου λοιπόν καλύπτονται από άλλους, άλλες οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με διακρίσεις λόγω ηθαγένειας και όχι άλλου τύπου. Στα όσα αναφέρθηκαν και τη διάκριση μεταξύ πολιτών Σέγγεν και μη Σέγγεν. Πολύ ενδιαφέρον βέβαια. Αλλά ίσως μπορεί να βρεθεί μια λύση. Στα σχόλια της Επιτροπής συζητήσαμε πολύ για το αν θα χρησιμοποιηθεί ο όρος μετανάστευση ε, εργαζόμενη σε κινητικότητα. Αλλά, όπως και να έχει, το, ότι, και έχοντας ακούσει διάφορα σχόλια, ο όρος αυτός μπορεί να αποτελέσει λόγο για παρερμηνίες. Αν πούμε μετανάστες ε, εργαζόμενοι, ενδέχεται να δώσουμε την εντύπωση ότι αναφερόμαστε εργαζόμενους από τρίτε χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει με κάποια διατύπωση που θα βρεθεί να ε, ξεκαθαρίσουμε ότι αφορά το εν λόγω νομοθέτημα μόνο τους ε, εργαζόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Συλλογικές αγωγέ. και παρατηρήσει του κύριου Κρίστινσεν θα πρέπει να συζητήσουμε βεβαίω. Πολύ ευχαριστώ να δω οποιαδήποτε άξια λύση. Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπήρξε αυτή η πρόταση και η σύσταση της Επιτροπής. Για τους διασυνοριακούς εργαζομένους, επίσης πρέπει να βρούμε λύση και περιμένω να ακούσω τι ιδέες μπορεί να έχετε, ώστε να μην αποκλειστούν, να μην αποκλειστεί κανείς. Για τα σχόλια της Προέδρου, ναι. Είναι πολλές φορές δύσκολη επιλογή. Δεν μπορεί να έχουμε ως στόχο να ε, αποστέλουμε εκατομμύρια εργαζομένων και να ανατρέπουμε τις δημογραφικές και πολιτισμικές δομές και αξίες. Ε, επί παραδείγματι, η Ρουμανία έχει γνωρίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εκατοντάδες ε, χιλιάδων ή χιλιάδες μόνο παιδιών εγκαταλελειμμένων στη Ρουμανία, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πέραν αυτού, αυτή η οδηγία έχει να κάνει με την ελευθερία της διακίνησης, δηλαδή την ε, απάλληψη των εμποδίων και φραγμών στην κινητικότητα. Δεν υποχρεώνει κανέναν να φύγει από τη χώρα του. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίζει, να έχει κανείς τη δυνατότητα για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια καλή ζωή, στην πατρίδα του πρώτα απ' όλα βεβαίως, αλλά ασφαλώς, ασφαλώς πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα της κινητικότητα, χωρίς βέβαια να μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι απλό το ζήτημα. Με το σχέδιο οδηγία προσπαθούμε πάντως, καθήκον μας είναι, να απαλείψουμε τα εμπόδια. διαπαντό. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 18 Σεπτεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Μετά εμείς ε, στις 17 Οκτωβρίου θα τις εξετάσουμε 5 Νοεμβρίου τις συμβαστικές και την ίδια μέρα μετά τα υπόλοιπα. Και έτσι θα μπορούσαμε υπό την προ... Ε, Λιθουανική Προεδρία να ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος αυτού. Να πάμε τώρα στο σημείο 10 και πάλι. Ο κύριος Κάζα έχει το λόγο και αυτό για να μας παρουσιάσει το σχέδιο του για την ΙΝΚΟ, την Επιτροπή για το Λιανικό Εμπόριο, Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης προς όφελος όλων των παραγόντων. Είναι από την ΙΝΚΟ, έκθεση πρωτοβουλίας. Έχετε το λόγο κύριε Κάζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα προωθώντα την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Ο τομέα του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει περίπου το 15% συνολική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλο ποσοστό νέων ατόμων. 29% όλων των επιχείρησεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται στον ε, τομέα αυτό. Περισσότερε από αυτέ είναι μικρομεσαίες επιχείρησει. Αυτή η γνωμοδότηση ε, καλεί να υποστηριχθούν περισσότερο καινοτόμες μεσαίες επιχειρήσεις ε, που ε, ανταποκρίνονται σε καινούργιες ανάγκε ανάγκες αγοράς και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους μικρούς λιανεμπόρους οι οποίοι ε, δυσκολεύονται περισσότερο να παρακολουθήσουν το ρυθμό που αλλάζει η τεχνολογία υπάρχουν ευκαιρίες ε, να ε, συμφιλιώσουμε ε, τις ανάγκες του λιανεμπορίου με, τις, με τη βελτίωση των προσόντων των νέων ατόμων. Η γνωμοδότηση συστήνει την ε, καλύτερη χρήση των υπαρχόντων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να υποστηριχθούν ε, συνεργασίες στο πλαίσιο του Εράσμους και άλλων προγραμμάτων. Η, επίσης, η ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασίων μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων πρέπει να υποστηριχθεί. Επίσης υπάρχει το θέμα της ε, αδήλωτης εργασίας ε, αποτελεί κοινωνικό κίνδυνο ε, γιατί αφορά χαμηλό, προσωπικό που αμείβεται πολύ χαμηλά, πολύ, λίγο και χωρίς κοινωνική προστασία. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Κομισιόν να έρθει σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους του λιανεμπορίου για αυτό το θέμα, με όλους τους παράγοντες. Θα συνεργαστώ με τους και ηγητές και τους συναδέλφους σε επόμενες εβδομάδες για να βελτιώσω το κείμενό μου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σορκάς και Μεταμπινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο κ. Κάσα, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πολύ σημαντικές για την ε, εσωτερική αγορά. Ο κ. Κοτσολίνο θα είναι ο υπεύθυνο από την ομάδα μας, μου έδωσε όμως ένα σημείωμα. Ε, αναφέρει ότι είναι ανοιχτό σε συνεργασία με τον κύριο Κάσα για να βελτιώσει το, το κείμενο παρόλο που δεν συμφωνεί πλήρως με τα όσα αναφέρει η έκθεση δεν γίνεται επαρκής ανάλυση ε, δεδομένου ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή σε αυτό το τομέα. Υφίσταται ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία οφείλονται στη συγκεκριμένη συγκυρία κρίσης. Αυτά δημιουργούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα για τους εργαζόμενους αλλά ε, και για τους τόπους τους οποίους λαμβάνει η χώρα η δραστηριότητα. Το λιανεμπόριο πλήττεται από μια διαδικασία ε, βαριάς αναδιάρθρωσης ε, που ε, στερεί την εργασία από πολλούς αλλά προκαλεί και σημαντικές ρήξεις στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Το λιανεμπόριο πλήττεται υπέρ των, και βγαίνουν δηλαδή κερδισμένες οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως σούπερ μάρκετ κλπ. Ε, παρόλο που το λιανεμπόριο στηρίζει και την οικονομική δραστηριότητα αλλά και την κοινωνία. Βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Ε, πέραν του τεράστιου ανταγωνισμού, άδικου ανταγωνισμού από πλευράς των μεγάλων σούπερ μάρκετ και των μεγάλων επιχειρήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, χειροτερεύουν πάρα πολύ οι εργασιακές συνθήκες. πλήττονται οι ίδιοι εργαζόμενοι αλλά και οι τους γιατί αλλάζουν τα ωράρια, ε, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται χιλιάδες από τους εργαζόμενους είναι υποχρεωμένοι χωρίς να το θέλουν να εργάζονται Σαββατοκύριακα πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε στην ΕΜΚΟ ότι πέρα από το εμπόριο και την ε, εσωτερική αγορά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από την ε, παραγωγικότητα και τα οικονομικά δικαιώματα ε, πρέπει να σκέφτεται και τους ανθρώπους. Όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα για να εξασφαλίσουμε την ευημερία των ατόμων. Πρέπει ε, οι επιχειρήσεις να, να είναι ε, στην υπηρεσία των εργαζομένων και όχι το αντίστροφο. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά δικαιώματα, η υγεία και ασφάλεια, τα ωράρια, τα μέγιστα ωράρια κλπ ο ανταγωνισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανισορροπίες, η αγορά, οι αγορές δεν είναι τέλειες, ε, δεν πρέπει να τις αγιοποιούμε, έχουν πάρα πολλές αδυναμίες και συνέπεια αυτών των αδυναμιών ε, είναι οι τεράστιες βλάβες, τεράστιες ζημίες τις οποίες ε, αναγκάζονται να φέρουν οι εργαζόμενοι. Θα συνεργαστούμε θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα ήθελα η Επιτροπή Απασχόληση όλοι μαζί, όλοι μαζί οι κοινοβουλευτικές ομάδες ε, να δώσουμε ε, τη δική μας οπτική γωνία ε, στην Επιτροπή ΜΚΟ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον κύριο Κρόιτσμαν, διότι ήταν σε άλλη Επιτροπή. Σήμερα διαβάζω λοιπόν τις σημειώσεις του κυρίου. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης και ε, για το λιανικό εμπόριο και για την αλυσίδα ε, προμήθειας μεταξύ των ε, επιχειρήσεων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρήσεις τη δεδομένη οικονομικής κρίσης. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό και ε, στο ΑΕΠ 15% της απασχόλησης, ε, άρα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο οι επιχειρήσεις αυτές για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πολύ περισσότερο δε βοηθούν στην λειτουργία τη εσωτερική αγοράς και την εγκυρητά της προς τον καταναλωτή. Έχουν πάντως πληγεί σημαντικά και αυτή είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής πόλης, που είναι και οι περισσότερες μικρομεσαίες. Ευχαριστώ τον συντάκτη για τις προτάσεις του. Επικεντρώνεται, όπως είπαμε, κυρίως στις ε, μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και τις μικρομεσαίες πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα συμβατότητας ε, στο εργατικό δυναμικό και συνθήκες εργασίας, αλλά ταυτόχρονα, λέει ο κύριος Κρότσμαν, χρειάζεται υποστήριξη για τις καινοτόμες μικρομεσαίες εταιρείες, ε, επιχειρήσεις και θα ήθελε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις ε, μικρές, στα μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου, στα κέντρα των πόλεων, αλλά και στην Ήπεθρο που κινδυνεύουν ε, ε, από τα πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα. Πρέπει λοιπόν να μπορούν και κυρίως οι ηλικιωμένοι που ζουν στην Ήπεθρο να... Μήπως κάποιος συνάδελφος θα επιθυμίσω το λόγο. Όχι, δεν βλέπω κανένα. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το επιθυμεί βέβαια, θα έχει το λόγο, ναι ή όχι. Be very brief for the Commission. Uh, uh, Θα είμαι πολύ σύντομη. Ο τομέας του λιανεμπορίου είναι πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία, το έχουμε πει επανειλημμένως, αλλά μην ξεχνάμε ε, επίσης και το γεγονός ότι ε, προσφέρει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Οι προτάσεις της ε, Κομισιόν λοιπόν είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικές. Ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα όλων των παραγόντων και του καταναλωτή και των λιανεμπόρων και των εργαζομένων. Θέλουμε να βελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια σε αυτό το ζήτημα. Το Συμβούλιο Εμπορίου για τα προσόντα, το, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κάσα, ήδη έτοιμασε την πρώτη του έκθεση τον Ιούλιο, θα συνεχίσει να δουλεύει. Η, η Συμμαχία των εργαζομένων σε μαθητεία επίσης έχει ε, ρόλο. Συνεπώς το σχέδιό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω θα εφαρμοστεί ε, με πολύ μεγάλο όφελος. Ε, η, το λιανεμπόριο λοιπόν έχει σχέση με θέσεις εργασίας αλλά και με μικρόμεσες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε δράσεις και για αυτές και η Κομισιόν θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές. Αυτά. Ο εις πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Συμφωνώ ότι η οικονομική κρίση έχει σε πολλές περιοχές της Ευρώπης οδηγήσει και σε κοινωνική κρίση. Και άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε βελτίωση των συνθήκων για τους εργαζομένους. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Μπίνιεν, υποφέρουν από την οικονομική δυσπραγία. Όπως προτείνει και ο κύριος Μπίνιαν και για τους και με τις ιδέες αυτές για τη βελτίωση των συνθήκων ε, για τους εργαζομένους στα εμπορικά κέντρα. Θα τα κοιτάξω πολύ προσεκτικά. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και τη συνεργασία για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα μάλλον να πούμε με ψηφιακές υπογραφές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στα αγγλικά 10 10 Σεπτεμβρίου Α, εντάξει 10 Σεπτεμβρίου Συμμάλλον σε όλες τις γλώσσες 25-26 Σεπτεμβρίου θα το εξετάσουμε ψηφοφορία 17 Οκτωβρίου μαζί με την εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών και η Επιτροπή ΙΜΚΟ δεν θα ψηφίσει τις 5 Νοεμβρίου. Πάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Βερονίκα, έχει το λόγο για την εξέταση των τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότησης για την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή για το εξάμεινο το ευρωπαϊκό για την εξάρτηση θεών μαζί και με τις προτεραιότητες για το 2013. Η έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, 88 τροπολογίες ε, που οι 88 τροπολογίες που διαθέτουμε θα βελτιώσουν το κείμενο. Οι συνάλφοι γνωρίζουν ότι το πρόβλημα που έχουμε πάντοτε είναι ο, ο περιορισμός ε, στο μήκος, ε, στο μέγεθος ε, Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ συνοπτικοί. Με τις 88 αυτές τροπολογίες νομίζω ότι η γνωμοδότηση θα διευρυνθεί και θα γίνει ε, ε, πιο πλήρης. Να αναφερθώ αρχικά στα πιο σημαντικά στοιχεία που θα θέλαμε να προσθεθούν στην έκθεση. Στρατηγική 2020, έχουμε μια σειρά τροπολογιών για αυτήν σχεδόν όλες από την συνάδελφο Κορνίλιεσεν που ε, αναφέρουν δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Σίγουρα ε, συμμερίζομαι αυτή την ανάγκη. Δέχομαι αυτές τις τροπολογίες. Μετά, απασχόληση των νέων είναι προτεραιότητα για την οποία έχουμε τροπολογίες επίσης. Έχουμε μία τροπολογία για τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων είναι από την κυρία Ζαλοβίσκα και με βρίσκει σύμφωνη. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες περί της μείωσης της φορολογίας της απασχόλησης. Αυτές οι τροπολογίες θεωρούν ότι αυτό είναι ένα μέτρο για, θα ήταν ένα μέτρο για την αύξηση της απασχόλησης. Συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα. Αλλά δεν πιστεύω ότι ε, θα έπρεπε εμεί να τοποθετηθούμε επί του πώς ε, θα αντισταθμιστεί αυτή η μείωση. Κάθε κράτος μέλος ε, θα πάρει τι δικέ του αποφάσει σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε με του κοιόδη. Ως ε, παράδειγμα θα μπορούσαμε να θέσουμε την εναλλακτική των περιβαλλοντικών φόρων όταν είναι ε, απαραίτητη. Μετά γίνεται λόγος για την ασφάλεια και την ελαστικότητα, την ευελιξία στις ε, εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει αυτές οι μεταρρυθμίσεις να περιλαμβάνουν την κατάλληλη ευελιξία για να είναι ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Όμως, το κριτήριο της ευελιξίας θα πρέπει να συμβαδίζει με τα κριτήρια της κοινωνικής οικονομίας αγοράς διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας. Ναι λοιπόν στην ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική προστασία. Τα τροπολογίες για τις δυνατότητες της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης από τον πράσινο τομέα, των, τομέα της πράσινης οικονομίας και για την, για τις, ε, την ανάγκη να επενδύσουμε στους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα. Και εδώ είναι καλές τροπολογίες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, τα οποία δεν θα σε αναφέρω πολλές λεπτομέρειες. Κάποιες τροπολογίες, οι οποίες μπορούμε αμέσω να υποστηρίξουμε, ενώ κάποιες άλλες θα τις λάβω υπόψη στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που θα προτείνω. Για παράδειγμα, πρόθεση της ποιότητας εργασίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μείωση της φτώχειας των εργαζομένων, συμφιλίωση της εργασιακής με την οικογενειακή ζωή, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των ε, ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν τελικά στην έκθεση. Επίσης γίνεται λόγος και για τους μακροχρόνιους άνεργους με μια σειρά τροπολογιών για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Επίσης γίνεται πολλής λόγους για την αργία των νέων, αλλά ε, θα πρέπει σίγουρα να συμπεριλάβουμε και τους ε, μακροχρόνια ανέργους. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες ε, δεν, καταλαβαίνω πολύ καλά, είναι δική μας αρμοδιότητα, αρμοδιότητα της ΕΚΟΝ η γραμματεία και σε συνεργασία με την πρόεδρο θα μας ενημερώσουν για το ποιε τροπολογίες είναι πιο πολύ αρμοδιότητα της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και ποιε είναι δικέ μας προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο μισθό, τον κατώτατο μισθό, Καλό είναι να το σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε με τον το αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο κείμενο να μιλήσουμε για τον το Παρόλο που δεν διαφωνούμε με την ιδέα. Για το Γιούρες. Αναφέρομαι κυρίως στον Σέρχιο Γουτέρες που λέει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του δικτύου EURES. Συμφωνώ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει το ρόλο αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να μιλήσουμε εδώ για το ρόλο του Γιούρες ως ε, διαμεσολαβητή για εργασιακά θέματα. Μετά, νέοι και κινητικότητα. Ε, κάποιοι θεωρούν ότι οι νέοι που μεταναστεύουν για να βρουν ε, ευκαιρίες σε άλλες χώρες είναι προβληματικό φαινόμενο. Ε, διότι χώρες όπως η δική μου χάνουν πολλά ταλέντα και μυαλά. Όμως να πούμε ότι είναι και αρνητικό φαινόμενο πρέπει να το δούμε θετικά. Είναι ανάγκη σε ορισμένες χώρες. Οι νέοι πρέπει να βρουν θέση, πρέπει να βρουν δουλειά. Αν δεν μπορούν να βρουν δουλειά στη χώρα τους, θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Μετά γίνεται λόγος για τον αυτόματο σταθεροποιητή. Τροπολογία της Προέδρου και του Σέρχιο Γκουτιέρες δύο τροπολογίε συγκεκριμένα που μου ζητούν η Κομισιόν να υποβάλει πράσινη βίβλο για την δημιουργία ε, επιδόματος ανεργίας για την Ευρωζώνη που θα λειτουργεί ω αυτόματος σταθεροποιητής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αλλά ίσως θα έπρεπε να το δούμε πιο προσεκτικά, ίσως μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί αυτό ε, σε μια τέτοιου είδου νομοδότηση όπως αυτή εδώ, παρόλο που δεν διαφωνούμε. Σήμερα το απόγευμα οι σκιώδες ηγητές θα πάρουν ήδη συμβαστικές προτάσεις και ημερομηνίες, ενδεχομένε ημερομηνίες για να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Γκουτήρες Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σημαντικό είναι, σημαντική είναι αυτή η στιγμή που τώρα συζητάμε για την έκθεση και επίσης ε, για τις τροπολογίες πέρα από τη συγκεκριμένη συζήτηση τώρα σχετικά με συγκεκριμένα θέματα εδώ που βλέπουμε διάφορες ομάδες με τις τροπολογίες και όπως τα αναφέρει η ίδια η έκθεση, αλλά πρώτα απ' όλα δύο κενά. Πολύ σημαντικά. Το πρώτα η όλη διαδικασία με όλες τις ε, για την δημοκρατική διαδικασία που εμείς ζητάμε περισσότερη συμμετοχή και για το εξάμεινο αυτό το ευρωπαϊκό. Αλλά εδώ στην τελική φάση πριν από την επεξεργασία αυτών των εθνικών σχεδίων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το επόμενο μήνυμα αυτή η έκθεση για αυτά τα εθνικά σχέδια είναι τώρα που υιοθετούνται από το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικότερο το πολιτικό μήνυμα από την πρακτική χρησιμότητα της έκθεσης να το λάβουμε υπόψη μας για να ασκήσουμε κριτική. Γιατί διαφορετικά θα είναι ψεύτικη δημοκρατία και θα πρέπει να το δούμε ανοιχτά, καθαρά. Δεύτερο τώρα, περισσότερη συμμετοχή από πλευράς Εθνικών Κοινοβουλίου είδαμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών βλέπουμε ότι εδώ με τους κοινωνικούς εταίρους δεν τα κάνουν όπως θέλουν και στα δύο αυτοτομείς και εμείς θα πρέπει να μας ανησυχεί αυτό το θέμα για να βελτιώσουμε αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία αυτή και την όλη δημοκρατία και την αίσθηση περί ηθαγένειας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα μια τρομερή απογοήτευση σε αυτές τις πολιτικές που αναπτύσσονται στα εθνικά σχέδια μεταρρύθμισης. Υπάρχει κάτι το λανθάνων ε, που κρύβεται στα διάφορα σχέδια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απογοήτευση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, έλαβε υπόψη της ε, την έκθεσή μας του Φεβρουαρίου που εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο. Όχι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε και κριτική και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, να το διορθώσουμε και ακόμα μια μικροανταλλαγή με αυτά τα προβλήματα, με τα προγράμματα ας πούμε προσοχής και περισσότερη ε, ευληγησία στο έλλειμμα και για τη μείωση του με μεγαλύτερη πίεση των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων που βάσει των εθνικών προγραμμάτων αυτών μεταρρυθμίσεων ε, έχουν να κάνουν με το κοινωνικό μας ε, πρόγραμμα κοινωνικό μας πρότυπο και ακόμα για τις ε, συντάξεις κλπ. που η Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει στόχους ε, μεσοπρόθεσμα, βραχυπόθεσμα, να δει πώς έχουν αυτά τα συστήματα, τα εργασιακά, τα συνταξιδοτικά και στα κάτι μελη τα περισσότερα και μερικές φορές ε, πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη χωρίς τον κοινωνικό διάλογο και την σεβασμό το δημοκρατικό και υπάρχει μια μικρό αλλαγή βέβαια σε αυτή την πολιτική και οι πολιτικές ομάδες ε, εδώ στην έκθεση όπως ε, υποβάλαμε διάφορες ε, τροπολογίες για καλύτερες συμβαστικές λύσεις γιατί χρειάζεται ένας κοινό παρόμοιος παρονομαστής αυτή την αλλαγή λοιπόν στις οικονομικές στρατηγικής σε όλα αυτά που είπαμε το Φεβρουάριο αλλά και πολλή ανησυχία γιατί γίνεται σε θέματα ακριβώς απασχόλησης είπαμε ναι ότι χρειάζεται παροτρυσή με πολιτική κατάλληλη. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης με κοινού παρονομαστές ασφαλείας και ποιότητας και για να ξεφύγει κανείς από όλα αυτά χωρίς μεγάλες διαφορές και αποκλήσεις και όλα αυτά δεν θα βοηθήσουν στο να ξεφύγουμε από την κρίση. Και ακόμα μια ανησυχία όχι μόνο για τους νέους αλλά χρειάζεται και για αυτούς που είναι μακρόχρονα άνεργοι. Θα πρέπει να το προσέξουμε και τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης πέρα από τώρα ε, θέλω να μας πούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι τα χειρότερα πέρασαν. Όχι όμως ε, δεν είναι αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται, ότι υπάρχει επιπλέον ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ε, ότι όλα αυτά θα ισχύουν μακροπρόθεσμα. Και ακόμα εμείς ε, την οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές, ε, εμείς μέσω τροπολογιών κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την περίφημη ανταγωνιστικότητα για να δούμε την έννοια αυτή, την ευρωπαϊκή οικονομία μας, πώς θα είναι περισσότερο ανταγωνιστική. Και θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για μια δήλωση του όλη Ρεν αυτό το καλοκαίρι που είναι αρμόδιο θέματα οικονομικά. Ζητούσε από την Ισπανία, α πούμε, από τη χώρα μου, ότι θα πρέπει 15 με 30% θα πρέπει να μειώσουμε το εργασιακό κόστος. Έτσι ακόμα περισσότερο να μειώσουμε τους μισθούς ε, ακόμη περισσότερο από ό,τι έγινε σε άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει φτώχεια και μείωση της κατανάλωσης και έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από την κρίση. Μας βοηθίζει ακόμα περισσότερο μέσω πρόθεσμα σε κρίση. Και ακόμα κάτι τελευταίο για την κινητικότητα. Είναι πολύ σημαντικές πολλές τροπολογίες ε, από τις διάφορες ομάδες που αναφέρουν το θέμα αυτό. Εδώ συμφωνώ εγώ και από αυτά που πρέπει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κοινωτικότητα όχι μόνο των κεφαλαίων αλλά και των εργαζομένων και αυτό που δημιουργήσαμε μέσω των διαφόρων εργαλείων ακριβώς είναι να διευκολύνουμε αυτή την κινητικότητα διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο και αυτή την κρίση την οικονομική που συμβαίνει σε πολλές χώρες είναι η διάθεση πραγματική να είναι κανείς πρόθυμος να το κάνει και όχι να το κάνει πιεζόμενος και που ποθεί νέος και λιγότερο νέος να εγκαταλείψει το κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υπέρ της κοινωτικότητας, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει ε, την οικονομική εξορία να την ε, πολεμήσουμε. Αυτό που γίνεται είναι δύο πράγματα. Δηλαδή, αν έχει κανεί με τη διάθεσή του να κάνει αυτά ή όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει το εξή. Πρώτα απ' όλα να βελτιώσει αυτό το ενδιάμεση ε, την μεσολάβηση. Είναι πολλά κρατημέλη που ακριβώς υπογράφουν διμερείς συμφωνίες έτσι, για κινητικότητα μεταξύ των εργαζομένων και είναι τρομερά, τρομερά λυπηρό. Αυτή τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ζούμε, όπου προσπαθούμε να δούμε ε, τι γίνεται με το χρέος, με τις τράπεζες κτλ. Να δούμε σε ποιους φορτώνονται όλα αυτά και για την ασφάλεια τους, ε, για τις συντάξεις τους και όλα αυτά που μας έχουμε σαν κοινωνικό πρότυπο. Θα πρέπει λοιπόν να μας ε, ανησυχούν όλα αυτά. Και όπως λέει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ε, τώρα που ξεκινάμε να βγαίνουμε από το τούνελ της κρίσης θα πρέπει όμως να ανησυχούμε και ιδιαίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο με όλα αυτά να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες θα ξεφύγουμε αυτό και πού πάει μας οδηγεί αυτή η έξοδος έτσι για να μην ανησυχούμε ακόμα περισσότερο για διάφορα θέματα και θα ήθελα να τονίσω όλα αυτά ε, που πραγματικά απασχολούν και κάνουν να υποφέρουν πάρα πολύ περισσότεροι από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Εδώ το λόγο έχει τώρα η Μαρία Άρκιν. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται η συγγετρία. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Συμφωνώ με πολλές από τις συστάσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή σχέση εργασίας. Πολλά από τα θέματα που ήθελα να θίξω έχουν ήδη αναφερθεί. Θα είμαι πολύ σύντομη. Οι τροπολογίες μου στο πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε ε, και βέβαια με δεδομένη την Ευρώπη των 27 και την οικονομική κρίση που δεν πιστεύω το μεταξύ να έχει αλλάξει ε, η αναλογία επί του ΑΕΠ ε, στο χρέος ορισμένων κρατών όλο και αυξάνεται και άρα χρειάζεται η ευελιξία για τη δημοσιονομική προσαρμογή και πρέπει να κοιτάξουμε όχι απλώς την ανεργία, αλλά τη μακροπρόθεσμη ανεργία. Με χαρά ακούω επίσης ότι θα υποστηρίξει σε έναν βαθμό έστω προοδευτικά φορολογικά συστήματα, κλιμακωτά δηλαδή, και θέματα τα οποία μπορεί να είναι βέβαια των κρατών μελών. την, ε, έστω και αν είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μερών, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και βέβαια για τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των κρατών των γυναικών κτλ. Ε, το κόστος του εργασιακού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ξέρω ότι το ξανασυζητήσαμε, αλλά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχει να κάνει και με την καινοτομία και με την έρευνα, με την επάρκεια των πόρων, με τη χρηματοδότηση. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες τροπολογίες πολύ σύντομα. Συμφωνώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην επιτύχηση στόχων του 2020. Πολύ σωστό αυτό, όπως και η εξισορρόπηση των κοινωνικών στόχων και των μακροοικονομικών στόχων ο κίνδυνος της διαρροής διανοιών ή της, ανισορροπ... της ανισορροπής κατά... κατανομής και ανατροπής των ισορροπιών μεταξύ ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού ή δημογραφικών αναταραχών. Στη χώρα μου έχουμε ε, αναχώρηση 10 ανθρώπων κάθε μέρα από τη χώρα με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Όταν καταλαβαίνετε ότι σαν χώρα όλοι μας ξεπερνάμε μόνο κατά ένα εκατομμύριο τον πληθυσμό του Βερολίνου, δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Επίσης ε, μίλησα για το φορολογικό χώρο, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Τροπολογίες επίσης από ε, την κυρία Καστελόρ, από την κυρία Κορνέλισεν για την ε, δημοσιονομική προσαρμογή που θα πρέπει να συζητήσουμε και για τον κύριο Πιέτο τροπολογία 86 όπου γίνεται λόγος για τη δημοκρατική νομιμοποίηση που απαιτείται πλήρω να εξασφαλίσετε. Φυσικά συμφωνώ και θα παρακολουθήσω και εγώ αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Όχι, θα κάνω εγώ μερικέ παρατηρήσει πριν να δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια και την Επιτροπή, αν το επιθυμεί. Καταρχάς, επιμένουμε ως προς την τροπολογία παριθμών 8 τον πίνακα στόχων ιδιαίτερα, ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο συχνά επανέρχεται, αλλά ιδιαίτερα στο έτος αυτό και ιδιαίτερα στα δεδομένα της ε, κατάστασης, χρειάζεται να έχουμε αυτά τα μέσα ανάλυσης και εξέτασης της καταστάσεως. Γι' αυτό παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Για την δημοκρατική νομιμοποίηση. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία έπεται των αποφάσεων του Συμβουλίου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία. Και στη τελευταία ανάλυση μπορούμε έτσι να εξετάσουμε και πώς λήφθησαν οι αποφάσεις του Συμβούλιο πώς ε, αποφάσεις, οι προτάσεις δικές μας του πρώτου τριμήνου έχουν ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο και αντίστοιχα βέβαια και τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα διδάγματα που θέλουμε να αντλήσουμε για το επόμενη περίοδο. Άρα πιστεύω ότι είμαστε συνεπείς με τα όσα έχουμε προτείνει. Για τον ελάχιστο μισθό που προτείνει η συγκήτρια. η επιχειρηματολογία σας ε, για τον ελάχιστο μισθό και το επίδομα ανεργία είναι νομίζω ταυτόσιμη. Ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό, εάν δηλαδή πρέπει να έχει θέση μέσα στην γνωμοδότηση αυτή, αν, έχει, αν είναι εδώ η θέση της. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να το περιλάβουμε το θέμα του ελάχιστου μισθού στην παρούσα γνωμοδότηση, γιατί ξέρουμε ότι αποτελεί μεγάλο διακύβευμα στην ισορροπία και στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μεγάλων των ε, οικονομιών της Ευρώπης. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει μελετήσει και παρατηρήσει και έχει προβάλει επιχείρημα για τη διατήρηση μιας κάποιας ε, ελάχιστης έστω εσωτερικής ζήτησης την ανάγκη για εισαγωγή αυτού του ελάχιστου μισθού ή τη διαφύλαξή του όπου υπάρχει ε, και επίσης για, την, ε, για το επίδομα ανεργίας διαπιστώνω ότι δεν, είσαστε, δεν κατά της, της τροπολογίας απλώς διαρωτάστε εάν έχει θέση μέσα στη βρωμοδότησή σας ξεκινήσαμε το θέμα και με την ακρόαση και με το πιλωτικό σχέδιο που ζητούμε να αναπτυχθεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον ορισμό του μακροοικονομικού πλαισίου, του συνολικού μακροοικονομικού πλαισίου που θεωρούμε απαραίτητο και χρήσιμο για τις κοινωνικές ε, πολιτικές της Ένωσης. Και άρα εστιαζόμενοι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα νομίζω ότι ναι, έχει θέση αυτό το επίδομα ανεργίας να το συστήσουμε. Και χωρίς να θέλω να αναπτύξω όλε τις τροπολογίες που έχω καταθέσει, μια ακόμη παρατήρηση για τι συντάξει. Και τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Πως ε, το μέσον αυτό για την ε, κατάθεση ειδικέ αναχώρα ειδικών αναχώρα προτάσεων αποτελεί και ένα μέσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει υποδείξει στα κράτη-μέλη. Και είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά εφόσον αυτές οι περίφημες ε, συμβάσεις καινοτομία και ανταγωνιστικότητα τελικά υλοποιηθούν. Αλλά εάν θέλουμε η μεταρρύθμιση των συντάξεων του συνταξιδοτικού συστήματος στα κράτη-μέλη να πραγματοποιηθεί πράγματι, πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ του να λέμε στα κράτη-μέλη, κοιτάξτε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών σα και του ταξιδιωτικού συστήματο και του να του υποδεικνύουμε πώ ακριβώ θα γίνει αυτή η προσαρμογή. Ή του να του λέμε ότι δεν θα πρέπει να σέβονται του κοινωνικού εταίρου, την αυτονομία του, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, τι διαρθρώσει που υφίστανται. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι εκείνη η οποία θα λέει η μεταρρύθμιση θα φτάσει μέχρι, θα, σημαίνει εργασία μέχρι τα 27, κεφαλαιοποίηση και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να απευθύνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένων των συστάσεων που είδαμε πέρσι. Για δε το δημοσιονομικό, στην τροπολογία 36, λυπούμε που δεν λέει τίποτα για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω βεβαίω ότι το φορολογικό σύστημα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά τόσα και τόσα λέει η Επιτροπή για τόσα θέματα που δεν είναι αρμοδιότητά τη κοινοτικής αρμοδιότητας δηλαδή. Ε, στο γενικό αυτό πλαίσιο των καλών προσανατολισμών, γιατί να μην είναι σιωπηλή ω προς το θέμα της φορολογίας. Της φορολόγησης, με τις συνέπειες δε που έχει η φορολόγηση ως προς τα έσοδα των κρατών μελών, ως προς τις συνθήκες χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και Άρα λοιπόν ελπίζω ότι θα γίνει δεκτή η τροπολογία 36 και θα την ενσωματώσετε στη γνωμοδότή σας. Η Επιτροπή θέλει το, το λόγο όχι, πολύ καλά, κερδίσουμε και μερικά λεπτά. Η συγκεκριά και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα είπαν ε, οι ομιλητές. Νομίζω ότι θα πετύχουμε μια συμφωνία. Ελπίζω να το πετύχουμε. Να δώσουμε όμως ε, ένα μήνυμα καθαρό στην Επιτροπή και πρόκειται για μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΕΚΟ για να δούμε να εγκρίνουν τις τροπολογίες αυτή την ε, που θα υποβάλλουμε προσεχώς την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε για να εγκρίνουμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πέρα τώρα από αυτή την εργασία της συγγήτριας μαζί με τον σκιώδη εμείς θα εξετάσουμε τις βασικές προτάσεις 18 Σεπτεμβρίου που θα ψηφιστούν τότε και η Οικονομική και η Νομισματική Επιτροπή θα ψηφίσει 30 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε μαζί με την συγκεντρία στην Οικονομική Νομισματική Επιτροπή να δώσουμε αυτή την ισχυρή ένδειξη, δείγμα των προθέσεών μας και που ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη. Πάμε τώρα στο 14 σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τι θα δούμε εκεί τις τροπολογίες στην έκθεση του κυρίου Κόζα την νομοδότηση στην Επιτροπή Γυναικών για την κατάσταση των αναπήρων γυναικών και θα δώσουμε στον αντικαταστάτη του συγητή το λόγο. Η κυρία Μπάουερ, ε, πρόεδρε ευχαριστώ. Ο κύριος Κώσσα δυστυχώς δεν είναι σε θέση να έρθει στη συνεδρίαση με επιφόρτηση να παρουσιάσω την νομοδότησή του. Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Βέρτμαν για την εξαίρετη συνεργασία. Ε, υπογραμμίζει ο κύριος Κώσσα ότι αυτή η συνεργασία έχει τεράστια σημασία και στο θέμα αυτό αφιερώθηκε ολόκληρη ημερίδα συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα για την ουσία. 38 συνολικά τροπολογίε έχουν καταθέσει συνάδελφοι. Τροπολογίε οι οποίε επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αναγνώριση δηλαδή πλήρου ισότητα για τι γυναίκε με αναπηρίε. Και ιδιαίτερα υπογράμμιση τη συμβολή του σε κάθε τομέα της κοινωνικής, οικονομικής ζωής. Ο κ. Σκόσα επεξεργάζεται μια σειρά τροπολογιών ως προς τη διαφορά στις αμοιβέ, ως προς την ανάγκη για ίση αμοιβή για ίση εργασία, απαγορεύονται οι, και διακρίσεις. Τρίτον, ε, δεύτερον, ε, οι πολλαπλές διακρίσεις θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και για λόγους φίλου βεβαίως. Το ζήτημα της μητρότητας και της άδειας μητρότητας θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη προσοχή. Με την κυρία Κλειβέτη συμφωνεί ο κύριος Κος ε, για τα φορολογικά κίνητρα. Στις προτάσεις του κυρίου Χιούιτ και άλλων, Χάουιτ και άλλων ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις γυναίκες και κυρίως στις γυναίκες με αναπηρίες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σύμφωνος. Κύριε Σκούσα είναι και μέλος της διπλωματευτικής ομάδας για τον τριμερή διάλογο και επισημαίνει διαρκώς τα θέματα αυτά. Είναι ευγνώμων προς τον κύριο Κλειδέτη, ο κύριο Κώσα, ο οποίος υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη προσβασιμότητα στην ε, επικοινωνία και την πληροφόρηση οι γυναίκες με αναπηρίες θα πρέπει να την χάνουν καλύτερης προστασίας κατά των ε, στο, στον χώρο της γενετήσιας ζωής. Ιδιαίτερα οι γυναίκες που είναι ιδρυματοποιημένες θα πρέπει να την χάνουν ιδιαίτερη απόδειξη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η, η, ανατροπή... η αναστροφή του βάρους απόδειξη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κατανομή των ε, γονεϊκών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων επίσης. Το να αναθρέψει το παιδί τη μια γυναίκα με αναπηρία δεν πρέπει να αποτελεί ένα μακρινό όνειρο, πρέπει να καθίσταται δυνατόν. Αυτά κυρία Πρόεδρε, εν ολίγης. Κύριε Λιβέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα ρουμανικά ως ε, σκιώδης εισηγήτρια. Εστίασα στις πτυχές σχετικές με την εργασία. Μια και οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν να αντιμετωπίσουν τα συνήθη προβλήματα των άλλων γυναικών, αλλά και τα πρόσθετα δικά τους. είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά τους και να λαμβάνονται, να υπόψη η δυνατότητά τους να δουλέψουν, οι ικανότητες και τα προσόντα τους και όχι οι αναπηρίες τους. Αυτές οι γυναίκες παράγουν κοινωνική αξία. Έχω υποβάλει 16 τροπολογίες θέλοντας να υπογραμμίσω την ανάγκη να τις ενθαρρύνουμε να γίνονται επιχειρηματίες, να καταπολεμηθεί ε, το φαινόμενο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και να, διευκολυνθεί, να διευκολυνθούν να γίνουν μητέρες. Στις τροπολογίες μου αναφέρομαι επίσης στην, στην κοινωνική βοήθεια, στην βοήθεια σε θέματα υγείας, γιατί εκεί ειδικά για αυτές τις γυναίκες πρέπει ε, να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να τις συνδράμουμε περισσότερο από τις άλλες γυναίκες. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Από ό,τι κατάλαβα από την κυρία Μπάουερ, ο εισηγητής, ο κ. Κώσα, συμφωνεί με τις περισσότερες από τις τροπολογίες μου, αν όχι με όλες. Πρόκειται για κατηγορίες ανθρώπων που έχουν συνεχώς ανάγκη την ε, βοήθειά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πραγματικά καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Εισηγήτρια, μήπως θα επιθυμούσατε το λόγο. Κύριε Χάρκιν. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κώσα για αυτή την πολύ πλήρη έκθεση. Έχω υποβάλει τέσσερις τροπολογίες που σχετίζονται με το θέμα των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όχι μόνο ότι υφίστανται μεγαλύτερο αποκλεισμό, αλλά και ότι ε, βρίσκουν πιο δύσκολα εργασία. Και όταν βρίσκουν εργασία έχουν μεγαλύτερη οικονομική εξάρτηση, μικρότερους μισθούς κλπ. Επίσης μίλησα για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, και για τις κοινωνικούς βοηθ, βοηθούς. Ε, το θέμα της πολλαπλής διάκρισης στο οποίο αναφέρεται κύριε Καβέτη, επίσης το θέμα της παρενόχλησης των και της βίας εναντίον των γυναικών. Ο κ. Χάουιτ έχει επίσης μια εξαιρετική ε, τροπολογία για τα εγκλήματα μίσους σε σχέση με τις αναπηρίες. Σε, πρόσφατη, σε πρόσφατο συνέδριο το θέμα συζητήθηκε και με πολύ λύπη ακούσαμε σχόλια που έγιναν από ανθρώπους με αναπηρίες ε, για ε, τις προσβολές που ε, δέχονται στο χώρο εργασία και τις καταχρήσεις. Επίσης, τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη οριζόντια στην, στον τομέα της κατάρτισης και της παιδείας. Θα πρέπει όλα αυτά να συνοδευτούν από απτή ενίσχυση, όχι να μείνουν στα λόγια. Ε, κάτι που επίσης νομίζω δεν υπάρχει στο κείμενο είναι ε, η ε, αναφορά στην ανάγκη για ανεξαρτησία στη ζωή, για αυτονομία. Και μετά η τροπολογία για την σεξουαλική βία κλπ. το βάρος απόδειξης θα αναφέρεται στην τροπολογία του κ. Χιούιτ ότι θα πρέπει να βαρύνει ε, τον ε, κατηγορούμενο. Όμως αυτό δεν είναι δυνατόν σε όλα τα νομικά συστήματα, ιδιαίτερα δεν είναι δυνατόν στο σύστημα, στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Κυρία Μπάουερ, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Θα ενημερώσω τον κύριο Κώσσα Οι συμβαστικές τροπολογίες θα ψηφιστούν στις 18 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Γυναικών θα ψηφίσει στις 3 Οκτωβρίου. Σημείο 15. Δίνω το λόγο στον Φιλ για να παρουσιάσει τις 45 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο σχέδιο γνωμοδότησής του ε, που απευθύνεται στην Επιτροπή ΕΜΒΗ για την οικοκαινοτομία, θέση εργασία και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Thank you. Yes. Uh, I'd like to thank my... Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, επικοδομητικές τους προτάσεις. Είδαμε πολύ καλές τροπολογίες Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Προτάσεις, πολλές από αυτές μπορώ να τις δεχτώ και θα υποβάλω και κάποιες ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες τις επόμενες δύο μέρες. Το συντομότερο δυνατό, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούμε την γνωμοδότησή μας να την περιορίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο Προσπάθησα να είμαι πολύ σύντομος λοιπόν και επιρρεκτικός. Τώρα με τις τροπολογίες μπορούμε πραγματικά να τη διευρύνουμε λίγο. Καταρχήν συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το πώς η οικοκαινοτομία μπορεί να βοηθήσει την ε, επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Ε, επίσης, η ε, αύξηση της ενεργικής απόδοσης των κτίριων δεν ε, κάνει πράξη μόνο την οικοκαινοτομία, αλλά μας βοηθάει να πετύχουμε και αυτού τους στόχους. Ε, κάποιοι συνάδελφοι αναφέρονται στην εκπαίδευση, ε, την ανάπτυξη προσόντων, την κατάρτιση, για να εξασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθούν οι δυνατότητες πρόσληψης, η προσληψιμότητα μέσω της οικοκαινοτομίας. Θα συμπεριλάβω και αυτές τις προτάσεις. Πολλές από αυτές τις προτάσεις σχετίζονται με νέους με νέου που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασία. Μην ξεχνάμε όμως και τους ανθρώπους που είναι βρίσκονται στην αγορά εργασία και πρέπει να επανακαταρτιστούν ε, γιατί βρίσκονται σε κλάδους ε, που ε, χάνονται ή μειώνεται η οικονομική τους ισχύς και πρέπει να διαφοροποιήσουν τον κλάδο στον οποίο εργάζονται. η οικογενοτομία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ε, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων απασχόλησης. Αυτό είναι αυτή είναι η ουσία της γνωμοδότησής μας. Αλλά δημιουργεί και καινούριες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να αναζωογονήσει παραδοσιακούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τρόπους να καινούριου τρόπου να εργαστούν και να διευρύνουν τι δραστηριότητε του. Αυτό θα έχει θετική επίδραση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Θα το τονίσω αυτό. ορίζω, όπως είπα, τις προτάσεις των συναδέλφων. στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι θετικές προτάσεις αυτές, αποδεκτές. Προσπαθώ να διοργανώσω μια συνάντηση με τους κοιόδους ηγητές την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω βρει ακόμα την κατάλληλη την κατάλληλη ώρα. Δείξτε λίγη υπομονή. Θα προσπαθήσω για την επόμενη εβδομάδα. Αν όχι, θα πρέπει να συνεχίσουμε μέσω email. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ας συνεχίσω στα γερμανικά. Κύριος Σμπανιέν επεσήμανε ότι θα πρέπει να παραμείνει η διασύνδεση με τη στρατηγική 2020 και νομίζω ότι αυτό σε πολλές συζητήσει λησμονείται πολύ συχνά, παραμένει όμως πολύ σημαντικός στόχος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με νέε θέσει εργασία, αλλά όχι μόνο με αυτό. Έχουμε να κάνουμε και με την προσαρμογή των υφισταμένων θέσεων εργασία στι νέε συνθήκε. Εγώ έχω μαζί με τον κύριο Μπάνιν αλλά και στο δικό μου μονόνομα καταθέσει κάποιες τροπολογίες για τα θέματα της κατάρτισης, ε, μετεκπαίδευσης, της έρευνας που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και εν γέννη, φρονώ ότι η στοχοθέτηση δεν είναι πάντα η ίδια. Ε, είναι πάντα η ίδια, προβλήματα δεν νομίζω θα έχουμε ως προς την συνεργασία και την εξέβρεση κοινού πεδίου. Θα ήθελα ωστόσο να ρωτήσω, αν και θα ήταν καλό να ήταν παρόντες όλες οι συνάδελφοι, όταν έρθει η ώρα με τους μπορούμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κούντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Σκιώδη εισηγείται εκ μέρου των Δημοκρατών. Δεν θέλω να πω ότι είναι πολύ καλή έκθεση και συμβάλλει σημαντικά στι κοινωνικέ πτυχέ και την κοινοτομία. Η ομάδα μας καταθέτει αρκετές τροπολογίες, ορισμένες ήδη ε, εφήγησαν. Ιδιαίτερα προβλήματα εγώ δεν διαπιστώνω σε σχέση με τις τροπολογίες. Πολύ σύντομα θα ήθελα να συνοψίσω τις τροπολογίες μας. Ε, μία ανάπτυξη πέραν της πράσινης και εφιούς ανάπτυξης και κοινωνικά αηφόρο. Αυτή πρέπει να σωματώσουμε, σύμφωνα και με τη στρατηγική. Ε, Επίση πρέπει να υπογραμμιστεί η ευθύνη των κρατών μελών, γιατί βλέπω να δίδεται πιο πολύ έφαση στις ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έπρεπε να δώσουμε πιο πολύ έφαση στι ευθύνε των κρατών μελών. Το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την κατάρτιση διαβίου μάθηση, αναμόρφωση, επιμόρφωση και το καθεξής. Αναφερθήκατε στους νέους και την οικολογική καινοτομία που γεννάνε στις για τους νέους, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και μετακύληση θέσεων εργασίας από τους πιο παραδοσιακούς τομείς μακροπρόθεσμα στον χώρο της οικολογίας και του περιβάλλοντος και πρέπει γι' αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη πως ε, θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας για μη ειδικευμένο προσωπικό, όχι μόνο δηλαδή υψηλό επίπεδο δεξιότητες, αλλά και ανειδίκευτοι εργάτες θα είναι απαραίτητοι. Ε, αυτό με την πτυχή βέβαια της κοινωνικής ενσωμάτωσης και βεβαίως οι περαιτέρω εξελίξεις ε, θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή όπως η συμμετοχή των γυναικών στην κατάρτιση και διαβίου το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την διαφύλαξη ή διατήρηση των χώρων εργασίας, ε, στη θέση εργασίας των ανθρώπων αυτών και προσέλκυση νέων, τα κίνητρα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης, που δεν επαρκούν και βέβαια το, το ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο αλλά και το εθνικό θα πρέπει να αναπτυχθεί και με διασυνοριακές συνεργασίες και κοινά ε, έργα, κοινέ ε, ε, συμπράξεις μεταξύ διαφορών κρατών μελών και ιδρυμάτων τους. Ε, αν έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν σε μια συνεδρίαση σκιωδών συγητών, πολύ ευχαρίστω, ε, αλλά μια και δεν υπάρχουν και πολλά διαφιλονικούμενα ζήτηματα, αν τυχόν δεν υπάρχει και ο χρόνο, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούμε να τα αλλάξουμε απόψει. Αλλά είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Δεν ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Ο κύριο Μπάνεν έχει το λόγο. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χάσουμε άλλο χρόνο, να καθυστερήσουμε. Τα σχόλια που ακούσαμε ήταν πολύ επικοδομητικά. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα βρει σύμφωνα τουλάχιστον τις τρεις ομάδες που εκπροσωπούνται εδώ. Πρόεδρος, ωραία, θα εξετάσουμε το αποτέλεσμα. Στις 18 Σεπτεμβρίου να μας υποβάλλετε ε, τροπολογίες ε, την ίδια μέρα θα ψηφίσουμε και στις 25 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και στην κατόπιν στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αυτά, σημείο 16, διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. και 24η συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου χτες. Ο λόγος στην κυρία Μωρόν Σαρτιέ. Σαρτιέ. Πράγματι 24η συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου. Έχουμε άλλες δύο στο πρόγραμμα. Χτες καταρχήν επιβεβαιώσαμε την αποτέλεσμα αποφασιστικότητα της Επιτροπής ε, Απασχόλησης έτσι ώστε το 25% των πόρων του Ταμείου Συνοχής να κατευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ε, να ε, μην παρεμβληθεί το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, μας ενίσχυσε αλλά και οι δυο Πρόεδρος και εγώ υποστηριζόμαστε και από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου μας. Οπότε ε, δεν είμαστε απομονωμένες σε σχέση με την Επιτροπή Ρέτζη. Δεν θα τελειώσει ο διάλογος, δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις ε, αν δεν ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Δεύτερον, όπως μας ζητήσατε στην εντολή που μας δώσατε, υπερασπιζόμαστε την πρόταση το 20% των πόρων του Ταμείου Κοινωνικής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να ε, ε, κατευθυνθεί στην ε, ενεργεία. Συγγνώμη, στην καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν ξέρω αν η πρόεδρος έχει την ίδια εντύπωση, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι δείχνει αυτή η πρόταση να μπορεί να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο σε μια τελική διαπραγμάτευση. Όμως το πιο πολύ εστιάσαμε στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων χτες. Σας υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό νέων μεταξύ 16 και 28 ετών σε, στην ανεργία. Εκεί που ε, ε, οι νέοι μεταξύ 16 και 25, οι νέοι άνεργοι σε ηλικίες μεταξύ 16 και 25, όχι 16 και 28, ξεπερνούν το 25%. Εμείς είχαμε ζητήσει ε, οι να μπορούν να δοθούν σε νέους μέχρι και 30 ετών συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματούχων. δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην ηλικιακή ομάδα 25 με 30. Επίσης, Τρίτο μας αίτημα ήταν αυτή η πρωτοβουλία για την αμασχόληση των νέων να είναι διαθέσιμη στις περιοχές που έχουν ε, ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 18 με 25 άνω του 20%. Ε, εδώ έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι το Συμβούλιο δέχεται για τις περιοχές που έχουν ενεργεία άνω του 25% για νέους 18 με 25 ε, να διευρύνει την ηλικιακή ομάδα στα 30 μέχρι τα 30, από 18 μέχρι 30 ετών δηλαδή. Αυτό το δέχεται το Συμβούλιο. Αντιθέτως, αγωνιστήκαμε πολύ για το 25% που θέλουμε να μειωθεί στο 20%. Ασφαλώς και το 20% είναι αυθαίρετο, αλλά το 25% είναι εξίσου αυθαίρετο. Τα θέλαμε, τους είπαμε, να ε, λάβουμε ως σημείο αναφοράς ε, το μέσο όρο, που είναι 22,9%. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους ανέργους. Οπότε ζητούμε οι περιοχές που έχουν ανεργία των νέων άνω του 22,9% δηλαδή ανεργία νέων μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο αυτές οι περιοχές να μπορούν να υποφελθούν από την ε, πρωτοβουλία. Τώρα, το Συμβούλιο λέει δεν πρέπει ε, να απαξιώσουμε αυτήν την πρωτοβουλία. Εμείς αγωνιστήκαμε έτσι ώστε ε, να, εστιαστού, να εστιαστεί αυτή η πρωτοβουλία τα έτη 2014-2015. Απ' την άλλη μεριά όμως μας λέει το Συμβούλιο προσπαθείτε να διευρύνετε την ηλικιακή ομάδα στο 30 έτη, να ρίξετε το ποσοστό στο 22,9% κλπ. Όμως έχουμε τα στοιχεία του Eurostat για τις περιφέρειες οι οποίε βρίσκονται σε, με ποσοστό ανεργία από το 22,9% στο 25%. Δεν είχα χρόνο να ε, μετρήσω, αλλά στην πραγματικότητα δεν απαξιώνεται η ε, πρωτοβουλία. Είναι πολύ λίγες αυτές. Δεν ε, έκανα θρήσεις ακόμα, αλλά θα το κάνω, έτσι ώστε να στηρίξουμε με περισσότερα επιχειρήματα αυτό μας το αίτημα. για να ληφθεί υπόψη ο μέσο όρο ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, δύο ακόμα σχόλια. Από τη Δευτέρα ακούω, φτάνουν στα αυτιά μου φήμε, ότι η συνεδρίαση τη επιτροπή Προπολογισμών τη Δευτέρα δεν προέβλεψε για το 2014, δεν συμπεριέλαβε την ε, πρωτοβουλία απασχόληση των νέων για τον προπερισμό του 2014. Θα διασταυρώσουμε τις πληροφορίες μας. Αυτές είναι όμως οι πληροφορίες που έφτασαν στα δικά μου αυτιά. Με θέτει όμως σε αμηχανία αυτό. Επίσης, ε, ρώτησα το Συμβούλιο χτες ε, για το εξής. Εμείς προσπαθούμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι το κείμενο θα είναι σαφές, θα το κατανοούν οι πολίτες μας, θα είναι ακριβές, απλό κλπ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες που το 2012 ε, απέφυγαν την εφαρμή του κανόνα κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου. Έχουμε και αυτό να ρυθμίσουμε λοιπόν με το Συμβούλιο. Ελπίζω να ήμουν πλήρης και εμπεριστατωμένη. Σας, δίνω το, σας επιστρέφω το λόγο για να σχολιάσετε, Πρόεδρε. Ε, για ποια συνεδρίαση μιλήσατε τη Δευτέρα, μιλήσατε για τη δική μας Επιτροπή για τους Υπουργούς. Α, για, όχι για την Επιτροπή ε, Προπολογισμών, αλλά για τους Υπουργούς Προπολογισμού. Το Συμβούλιο Προπολογισμού δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω κάτι, καμιά πληροφορία σχετικά με αυτό. Δύο παρατηρήσεις να κάνω όμως. Πρώτη παρατήρηση τι κατακτήσαμε σε 30 χρόνια και βλέπουμε ότι το Συμβούλιο αυτό εξαρτάται από το 25% ανεργία σε μια περιοχή και όμως αυτό ισχύουν για μια σύμφωνη δεχόμενη με το Συμβούλιο. Εντάξει, δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να προσθέσω τώρα. Ενώ υπό την Προεδρία αυτή δεν θα γινόταν. Ε, για την εγγύηση για την νεολαία πετύχαμε στον κανονισμό αυτό μια αναφορά. Για μας ε, αποτελούσε ένα ε, σημείο δύσκολο να το πετύχουμε, να το πετύχαμε. Μήπως κάποιος θέλει κάτι να ξέρει, όχι, εντάξει, συγχαρτήρια στην Επιτροπή Διαπραγματεύσεων και εντάξει, μετά από το 20ο τριμερή διάλογο, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα συνθούμε, Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε τη μεσιά διάταξη και αν δεν έχει κανεί κάτι για τα διάφορα, τότε η επόμενη μα συνάντηση 18 Σεπτεμβρίου, κυρίε και κύριοι.